Good afternoon, everyone. you are willing to take Καλό σας απόγευμα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είναι εδώ μαζί μας ο, ο Dr. Μπαχίντο Μοέτη, ο Περιφερειακός Διευθυντής για την Αφρική της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας από την Ποτσουάνα. Είναι η πρώτη γυναίκα περιφερειακή διευθύντρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ε, είναι, έχει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το 1999 ε, άρχισε να εργάζεται στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και έχει διατελέσει ε, επικεφαλή σε μια σειρά από περιοχές. Αυτή η ανταλλαγή απόψε ήταν μια ευκαιρία να συζητήσουμε την υγεία στα πλαίσια των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα δώσουμε έμφαση στις μεταδοτικές ασθένειες και στις εκτάκτες, ε, στις, εξε, στις ε, επίγουσες περιπτώσεις υγείας. Είναι εδώ και εκπρόσωποι ε, βουλευτές από την Αφρική, είναι εδώ στα πλαίσια της Αφρικανικής Εβδομάδας, από το Παναφρικάνικο Κοινοβούλιο είναι εδώ κάποιοι εκπρόσωποι από το Κοινοβούλιο της Νιγηρίας, από το Μαρόκο και από την Τινησία, από το Κοινοβούλιο της Τινησίας. Ξέχασα κανέναν. Όχι. Ωραία. Καλώς ήρθατε εκ νέου και να, ξεκινήσουμε τη σημερινή συνάντηση. Βεβαίως θα ήθελα πρώτα να καλέσω την Δόκτωρ Μοέτη να πάρει το λόγο και να μοιραστεί μαζί μας κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθώς και τις εμπειρίες της σε αυτήν την πολύ σημαντική θέση την οποία έχει αναλάβει στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Αφρικανικής Ένωσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκονται εδώ ε, και βουλευτές ε, από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο αλλά και από μια σειρά χωρών της Αφρικής. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που με καλέσατε πρώτα απ' όλα σε αυτή την Αφρικανική εβδομάδα για να έχουμε μια συζήτηση για την υγεία στην Αφρική. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα μεγαλύτερα ζητήματα υγείας, τα οποία για μας το μεγαλύτερο ζήτημα είναι οι μεταδοτικές ασθένειες. Ε, βεβαίως ε, έχουμε και υψηλά ποσοστά ε, θανάτων κατά την γέννηση των καροντοκετό ε, των μητέρων. Ε, οι χρόνιες ασθένειες επίσης έχουν εξαπλωθεί. η Ήπειρός μας, η ευρύτερη περιφέρεια, ε, έχει να αντιμετωπίσει ε, ένα διπλό βάρος ασθενειών ε, και χρειάζονται πολλές και επικίνδυνες απαντήσεις για τη διαχείριση αυτών των φαινομένων. Είναι λοιπόν χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις για να δούμε πώς με τις χώρες της Ευρωπαϊκές, με τις χώρες της Αφρικής μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτή τη διπλή επιβάρυνση από ασθένειες. Αυτή η συζήτηση λαμβάνει η χώρα στα πλαίσια των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη είχαμε αυτήν, αυτό το πλαίσιο το οποίο εμπνέει, εμπνέει την Αφρική, ε, δημιουργούνται δυνατότητες, ε, έχουμε, δίνεται μεγάλη, πολύ μεγάλη τρέφαση προς το παρελθόν ε, στην υγεία, στην Αφρικανική Ήπειρο. θέλουμε να εξασφαλίσουμε βεβαίως υγιή διαβίωση, ε, και αυτό είναι στην καρδιά της προσπάθειάς μας. Η υγεία ε, σχετίζεται με όλους τους άλλους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Πολλοί από τους στόχους αυτούς ε, εξαρτώνται από την υγεία και επηρεάζονται από την υγεία. Η υγεία θα μπορούσε λοιπόν να συνεισφέρει και για την επίτευξη των άλλων στόχων. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να προωθήσουμε και να θεσπίσουμε μηχανισμούς για να εργαστούμε πολυτομεακά, πολυτομεακή δράση όπως λέμε, ε, σε διάφορους τομείς πολιτικής. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται σε άλλους τομείς συνεισφέρουν ή τουλάχιστον ε, δεν επιδεινώνουν ε, την κατάσταση της υγείας. Είναι κάπως διαφορετική δηλαδή η προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν. Έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Ελπίζω να βλέπετε τις διαφάνειες και αυτές οι επενδύσεις στην Αφρική έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουμε σημαντική μείωση στην παιδική θνησιμότητα, ε, παρότι η περιοχή της Αφρικής ε, έχει πολύ ψηλά ποσοστά AIDS, ε, έχουν μειωθεί τα κρούσματα, τα νέα κρούσματα και αυτό οφείλεται, ε, αυτό έχει να κάνει, μάλλον, μάλλον τα νέα κρούσματα είχαμε και για το AIDS και για την ελονοσία τα οποία όμω μειώνονται ακριβώ χάρη στην προσπάθεια που γίνεται στα πλαίσια τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίση, υπάρχουν τεράστιε ευκαιρίε ε, με βάση τι νέε δεσμεύσει από τι αρχέ, ε, τι αυξημένε επενδύσει στον τομέα τη υγεία, παρότι βεβαίω αυτέ οι επενδύσει δεν έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο για να μπορέσουν περισσότερε χώρε ε, να παρουσιάσουν ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών υγιεινής να υπάρχει απαραίτητη πρόληψη για να μπορέσουν να αντιστραφούν τα ποσοστά θνησιμότητας. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες, η έρευνα, η τεχνολογία ε, οδηγεί σε νέα εργαλεία, σε νέες μεθόδους εργασίας που θα πρέπει οι χώρες της Αφρικής να εντάξουν στα προγράμματά τους για να μπορέσει η περίθαλψη αλλά και η πρόληψη να είναι πιο αποτελεσματική. Έχουμε πολλούς, ε, έναν πολύ νεανικό πληθυσμό ε, και οι νέοι ε, είναι δημιουργικοί, προσαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα στην τεχνολογία. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσει, αλλά και ο ιδιωτικό τομέα πολύ γρήγορα να ενσωματώσουν ε, αυτά, αυτές τις νέες τεχνολογίες. Ο κόσμος μας ε, διέπεται από όλο και μεγαλύτερη διασύνδεση. Είχαμε μια τεράστια επένδυση σε όλο τον κόσμο στο μέρο τη πρόληψη, μόνο και μόνο για τρει χώρε τη Αφρική πριν από λίγο καιρό. Ε, όταν εμφανίζονται μεταβατικέ ασθένειε, υπάρχει δηλαδή αντίδραση παγκοσμίω. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό, ότι ο κόσμο μα είναι ένα, είναι ενιαίο και ε, είναι όλο και πιο ε, αλλη, Αυτό συνέβη λοιπόν με την περίπτωση, του έμπολα, ε, όπου η αντίδραση ήταν άμεση, ε, έτσι ώστε να μην εξελιχθεί σε πανδημία αυτά τα κρούσματα που λοιπόν, εμφανίστηκαν στι τρει χώρε τη Αφρική, της τα κρούσματα έμπολα. Θα αναφερθώ εν συντομία στις βασικές ασθένειες που ε, πλήττουν τον αφρικανικό πληθυσμό σήμερα. Το AIDS, πρώτα απ' όλα, βεβαίως γνωρίζουμε ότι η περιοχή της Αφρικής είναι πλέον ε, ε ενδιαφερόμενη περιοχή Μιλάμε για 5 εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ε, έχουν AIDS ε, και είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται να το αντιμετωπίσουμε. Μόλις πέρυσι 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι ε, μολύνθηκαν από το AIDS και έχουν και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος βεβαίως ε, για να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβαση στα, σε, σε θεραπεία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ε, βλέπουμε ανθρώπους δηλαδή να πεθαίνουν από AIDS ε, τις ίδιες εικόνες που βλέπαμε και πριν εμφανιστεί η θεραπεία. Έχει μειωθεί η πρόοδος λοιπόν σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την Ήπειρο για την καταπολέμηση του AIDS ε, αλλά οι χώρες της Δυτικής Αφρικής, της Κεντρικής Αφρικής, εκεί που η, αυτή η επιδημία δεν είχε τόσο, ε, δεν ήταν τόσο διαδεδομένη, εκεί λοιπόν είναι πιο αργή η πρόοδος, διότι υπάρχει ένα συγκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος υγείας, όταν ε, οι πρωτοβουλίες μας φτάσαν εκεί για να αυξηθεί η πρόσβαση στην θεραπεία, ε, έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι ε, δεν φτάνουν οι γιατροί. Έπρεπε λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα και σε μια νοσοκόμα να ε, περιθάλψει έναν ε, φορέα του ιού. Έχει γίνει μια προσπάθεια Πάλι τώρα στις χώρες της Κεντρικής Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής. Υπάρχει ένα επίγον πρόγραμμα ε, για την επιτάχυνση της προόδου, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα κενά. Είμαστε πάντως αισιόδοξοι. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο στόχος του να πάψει το AIDS να είναι ε, ζήτημα δημόσιας υγείας ε, μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή της Αφρικής. Ε, υπάρχει κλιμάκωση της πρόσβασης στη θεραπεία. Ε, έχουν γίνει επενδύσεις και από το Παγκόσμιο Ταμείο, από το πρόγραμμα ΠΕΦΑ των ΗΠΑ. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε σωστή οδό έτσι ώστε 20 εκατομμύρια άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη θεραπεία αυτό που θα πρέπει να συμβεί βέβαια είναι οι εθνικές κυβερνήσεις να επενδύσουν και δικούς τους πόρους ε, για τα προγράμματα θεραπείας. Ε, η αποκέντρωση δεν έχει συμβεί ακόμα, παρότι έχει μειωθεί το ποσοστό μόλυνσης, ε, εξακολουθεί να υπάρχει αύξηση στα νέα κορίτσια Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν δηλαδή διακρίση μεταξύ των φίλων, οι νέε γυναίκε ε, που έχουν ε, σεξουαλικέ σχέσει με ε, γυραιότερου άντρε, οι σχέσει εξουσία που υπάρχουν, ένα κώδικα σιωπή όπου που, μια επιβαλόμενη σιωπή, όλα αυτά είναι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς και το υψηλό ποσοστό μόλυνσης στα νέα κορίτσια. Υπάρχουν κάποιες, κάποιοι πληθυσμοί κλειδιά στην περιοχή, ε, οι ομοφιλόφιλοι άντρες, ή ε, τοξικομανείς. Ε. Ελπίζουμε πάντως, έχουμε, βλέπουμε εδώ ένα παιδί το οποίο περνάει από τεστ. Ε, υπάρχει μεγάλη αύξηση στην πρόληψη ε, για την τη μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο παιδί. Αυτό είναι μια θετική εμπειρία. Θα αναφερθώ τώρα εν συντομία στη φυματίωση και μια άλλη ασθένεια ε, που πλήττει δυσανάλογα πολύ την Αφρική. Περίπου 40% του παγκόσμιου πληθυσμού 25% του παγκόσμιου Παγκοσμίω, ε, σε ό,τι αφορά τη φυματίωση, προέρχεται από την Αφρική. Συχνά, επίσης, όσοι έχουν AIDS ε, είναι πιθανό να αναπτύξουν φυματίωση. Ε, η φυματίωση, άλλωστε, είναι ένα από του βασικούς ε, βασικές θανάτου φορέων AIDS. έχουν, έχει, έχει εμφανιστεί και μια φυματίωση που είναι ανθεκτική τα φάρμακα, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ότι τα φάρμακα αυτά ούτως ή είναι πολύ ακριβά, γνωρίζουμε ότι η φυματίωση, αναγνωρίζουμε μάλλον ότι η φυματίωση είναι άλλη μια ασθένεια που χρειάζεται πολυτομιακή προσέγγιση. Οι πιο ευάλωτες ομάδες ε, είναι ε, ε στην Νότια Αφρική, παραδείγματο χάρη όσοι εργάζονται στα ορυχεία, εκεί είχαμε πάρα πολλέ περιπτώσει φυματίωση Άνθρωποι που δουλεύουν εδώ και δεκαετίε. Ε, εκτεθειμένοι στη σκόνη, αυτοί που δουλεύουν επίσης στον τομέα των, της οικοδομής, άνθρωποι που είναι στη, στη φυλακή, ε, στα σοφρονιστήρια και εκεί λόγω των συνθήκων εντό των φυλακών είναι πολύ ευάλωτοι, ευάλωτοι πληθυσμιακές ομάδες. Ε, γίνεται μια προσπάθεια να αναπτύξουμε νέα εργαλεία για τη φυματίωση. Υπάρχει πρόοδος σε επίπεδο διάγνωσης, επίπεδο θεραπείας είναι πιο, πολύ πιο μικρή η διάρκεια της θεραπείας, μπορούμε πλέον να επιταχύνουμε ε, τις διαδικασίες αυτές. Είναι όμως εφικτό και επίσης ε, η φυματίωση να εκλείψει ως πρόβλημα για τη δημόσια υγεία έως το 2020 εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες επενδύσεις. Τα προγράμματα για την φυματίωση στην περιοχή έχουν ε, μια χρηματοδότηση τάξη του 40%. Είναι περιορισμένες υπηρεσίες που μπορούν να ε, παρα, να, να υπάρξουν. Έγινε μια συνάντηση στη Μόσχα την προηγούμενη εβδομάδα για την φυματίωση. Υπήρξε μια δήλωση, δήλωση τη Μόσχα με τη δέσμευση τη επιτάχυνση των εργασιών γύρω από τη φυματίωση και την ε, ιδέα να υπάρξει μια συζήτηση, μια διάσκεψη στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών ε, για τη φυματίωση, να αναγνωριστεί δηλαδή η διάσταση του προβλήματος και εδώ στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες. Ελπίζουμε να μπορέσουμε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να ενδιαφερθούν για το ζήτημα αυτό ε, και έτσι ώστε να υπάρξει η απαραίτητη χρηματοδότηση, ε, να γίνει η απαραίτητη δουλειά για τη φυματίωση, κάτι που δεν έχει συμβεί ως τώρα σε σχέση παραδείγματος χάρη με το AIDS. Θα πρέπει να συμμετέχουν βεβαίως και οι πολίτες ε, όπως για το AIDS υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχουν ακτιβιστέ ε, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ρίξουν τι τιμέ των φαρμάκων που κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει με τη φυματίωση. Τώρα η Ελλονοσία Ε, η Ποσαχάρη Αφρική είναι έτσι, η έδρα της Ελλονοσία παγκοσμίω. Έχουμε περίπου ε, είχαμε περίπου 395 νεκρούς ε, και εδώ έχει σημειωθεί πρόοδος ε, για τη μείωση των περιπτώσεων Κατά τη διάρκεια το, της περίοδου της ανάπτυξης των στόχων της χιλιετίας ε, υπήρξαν προγράμματα σε μια σειρά από χώρες, ε, επενδύσεις μέσω του Παγκόσμιου, του Παγκόσμιου Ταμείου και άλλες ε, πρωτοβουλίες χρηματοδότησης. Έτσι λοιπόν ο αριθμός των περιπτώσεων ελονοσίας μειώθηκε κατά 6,8 εκατομμύρια. 6,8 εκατομμύρια λιγότεροι θάνατοι και 633 εκατομμύρια λιγότερες, ε, λιγότερα κρούσματα, λιγότερες ε, λιγότεροι ασθενεί. Ε, είχαμε επίσης και νέες τεχνολογίες, ε, μία αύξηση των δοκιμών στα παιδιά, των τεστ στα παιδιά, διότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην ελονοσία και ελπίζουμε πραγματικά ότι με μια σειρά εργαλεία, με τον ντομοκτώνα, ε, την γρήγορη θεραπεία, διάγνωση και θεραπεία, υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα που δοκιμάζει ένα εμβόλιο κατά της ελονοσίας που θα προσφέρει ε, μια έστω και μερική ε, προστασία. Με αυτά λοιπόν τα μέσα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να μειώσουμε σημαντικά τα, τις περιπτώσεις ελονοσίας. Ε, τέλος, σε ό,τι αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες, θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπικές ασθένειες που προέρχονται από την Ασία ασθένειες ε, που έχουν να κάνουν με τον ύπνο, ελεφαντίαση, ε, ασθένειες ε, που επηρεάζουν κυρίως κοινότητες χαμηλών εισοδημάτων στην ύπεθρο, που παραλύουν τη δυνατότητα των ανθρώπων να εργαστούν, να παράγουν τρόφιμα και ουσιαστικά δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο φτώχειας. Δηλαδή ήδη φτωχέ κοινότητε ε, γίνονται φτωχότερε εξαιτία αυτών των ασθενειών. Ε, το 2012 έγινε μια διάσκεψη στο Λονδίνο όπου η διεθνή κοινότητα, οι κυβερνήσει, οι κοινωνίε των πολιτών, ε, διάφορες φιλανθρωπικέ οργανώσεις αποφάσισαν να επιταχύνουν τι εργασίε και τι επενδύσεις για αυτές τις παραμελημένε τροπικές ασθένειε, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκριζωθούν τουλάχιστον κάποιες από αυτές και να μπορέσουν αυτές οι κοινότητες να απαλλαγούν ε, από τις ασθένειες αυτές που χρειάστηκε ε, να τους χορηγηθούν μαζικά φάρμακα για να ελεγχθεί η ασθένεια. Το Τογκό ήταν η πρώτη χώρα στη Δυτική Αφρική ε, που κατάργησε, που κρίζωσε την λεμφατική με ελαφατική ασθένεια και είναι και άλλε χώρε που είναι κοντά, όπω το Μαλάουι. Προσπαθούμε λοιπόν να συνεργαστούμε και με τη φαρμακοβιομηχανία που ε, δορίζει κάποια φάρμακα έτσι ώστε να υπάρξουν κάποια μαζικά προγράμματα πρόληψη για να μπορέσουν να κρυζώσουμε αυτέ τι ασθένειε και να μην χρειάζεται πλέον να επενδύσουμε εκεί. Είναι μια καλή επένδυση αυτή. Ε, θεωρούμε ότι 50 cents ανά άτομο το χρόνο είναι όσο χρειάζεται, όσα χρήματα χρειάζονται για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτές τις ασθένειες. Είναι λοιπόν μια καλή επένδυση. Η περιφέρειά μας ε, ε, συχνά παρουσιάζει επιδημίες και κρούσματα μεταδόσιμων ασθενειών, μεταδοτικών ασθενειών. Αναφέρθηκα προηγουμένως στα κρούσματα έμπολα. Ε, νομίζω ότι αυτό έχει ε, ε δημιουργήσει μεγάλη ζημιά στη συλλογική, στο συλλογικό ψυχισμό των ανθρώπων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι απαραίτητε δυνατότητε για να εντοπίζονται αυτά τα κρούσματα έγκαιρα, να μην τα αφήνουμε να εξελίσσονται σε επιδημία. Ε, έχουμε περίπου 100 ε, γεγονότα δημόσιας υγείας ετησίως, γεγονότα το ονομάζουμε εμείς, Οπότε είναι συνεχής η προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπίσουμε. Ε, συνήθως έχουμε να κάνουμε με χολέρα, ε, έμπολα, ε, μενιγκίτιδα, κίτρινος πυρετός, ε, μια σειρά από τέτοιε ασθένειε. Είχαμε και μια πανούκλα, μια, ε, είχαμε την πανούκλα που πανίστηκε στη Μαδαγασκάρη πρόσφατα. Επίση υπάρχουν περιοχέ του κόσμου όπου εμφανίζονται κάποιες ασθένειες όπως στη Βόρεια Αφρική, στην Κεντρική Αφρική, ε, εκεί όπου υπάρχουν σειράκες στον Νότιο Σουδάν, όπου η δυνατότητα της δημόσιας υγείας να, ε, να λειτουργήσει είναι εντελώς ε, προβληματική, δηλαδή εμφανίζονται ακόμα και κρούσματα μαγουλάδων μαζικά επειδή δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ε, υπάρχει το θέμα της ε, ε μικροβιακής αντίστασης, αυτό είναι παγκόσμιο πρόβλημα επειδή υπάρχει μαζική χρήση αντιβιωτικών, αλλά όχι μόνο στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και στην, στο περιβάλλον, στην γεωργία και αυτό έχει επηρεάσει και τι περιβαλλοντικέ συνθήκε. Όλα αυτά αποτυπώνουν το γεγονό ότι το σύστημα τα υγεία στι χώρε αυτέ δεν είναι αρκετά στεναρά, δεν είναι αρκετά ισχυρά, δεν υπάρχουν αρκετέ εγκαταστάσει, αρκετό προσωπικό με τι κατάλληλε δεξιότητε, αρκετά εργαστήρια για να ε, εντοπίσουν και να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη κρουσμάτων ε, ακόμα και απλή, απλές διαδικασίες πρόληψης κάποιων ε, μολύνσεων ε, στο, είδα, στο, είδα, στο ίδρο παραδείγματος χάρη δεν λαμβάνουν χώρα και αυτό οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα. Όσο παγκόσμια οργάνωση υγείας αντιδρούμε με διάφορους τρόπους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ να βελτιώσουν τι δυνατότητε του. Λοιπόν, θεωρούμε ότι με αυτή την επιβάρυνση από τις ασθένειες, αλλά και με την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά διεθνείς επενδύσεις, αλλά και την αυξανόμενη δέσμευση από τις χώρες αυτές, ε, έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο, παραδείγματο χάρη για την κατάργηση, την εκρίζωση μάλλον της πολυομιελίτιδας έως το 2000 είχαμε πει, ε, και βλέπουμε ότι σε χώρες όπου υπάρχουν σειράξεις ένοπλες ε, ένα χρόνο αφότου ε, ε, γιορτάσαμε την εκρίζωση της πολυμελίτιδας εμφανίστηκε εκ νέου ε, και αυτό συμβαίνει και σε χώρες άλλες όπου υπάρχουν σειράξεις ε, στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και, και μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και με αρχές ασφαλείας που ποτέ, ποτέ πραγματικά ε, δεν φανταζόμουν μόνο ότι θα συμβεί αυτό. Να συνεργαζόμαστε καθημερινά με το στρατό, μπορούμε να πάμε εκεί, μπορούμε να πάμε να καθαρίσουμε, να παρέμβουμε, να, κάνουμε μια εκστρατεία ε, εμβολιασμού. Αναγκαζόμαστε ε, να μάθουμε νέους τρόπους ε, συνεργασίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τη βοήθειάς μας. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο AIDS, στην ελονοσία, στην φυματίωση. Ε, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε αυτές τις ασθένειες χρειάζονται ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας με επαρκή χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο ε, για να μην χρειάζονται οι άνθρωποι να πληρώνουν στο σημείο περίθαλψης όταν βλέπουν τον γιατρό αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχουν κάποια συστήματα ασφάλειας με τους κατάλληλους πόρους να έχουν συγκεντρωθεί έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση και αυτοί και, και τα χαμηλά εισοδήματα ε, να, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε δηλαδή περαιτέρω ρόλο τη δημόσια υγεία στι χώρε αυτέ. Αυτό συνδέεται με την καθολική ε, ιατρική κάλυψη. Ε, αυτός είναι ο στόχος μας. Ε, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες ε, των πληθυσμών. Η Υπουργή Οργάνωση υγεία έχει δημιουργήσει μια έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για αυτήν την καθολική κάλυψη. Είχαμε μια προσέγγιση που βασιζόταν σε συγκεκριμένε ασθένειες και έχουμε καταλάβει πλέον ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αφορά και την πρόληψη και την περίθαλψη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα του πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα στα πλαίσια των διαφόρων προγραμμάτων και να τα επενδύσουμε και αυτά για την οικοδόμηση συστημάτων δημόσια υγεία στι χώρε. Ω μέρο αυτών που κάνουμε για να μπορέσουμε να εστιάσουμε, να αλλάξουμε την εστίαση, να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τι χώρες μας για να βελτιώσουν τα συστήματα υγείας τους, να, να τα ενισχύσουν. Σας δείχνω εδώ μια διαφάνεια, υπάρχει ένα δείκτη όπου προσπαθούμε να εκτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε την κάλυψη με ένα, κάποιων βασικών υπηρεσιών υγείας. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μεγάλη ε, Η χώρα που βλέπετε πάνω πάνω είναι η Αλγερία, όπου έχουμε περίπου, που φτάνει στο 80 και το, ο Νίγηρας που είναι κάτω-κάτω είναι στο 11 ε, σε ό,τι αφορά την κάλυψη. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι τεράστια διαφορά από το 80% στο 11% σε ό,τι αφορά τις χώρες ε, και τη δυνατότητά τους να παράσουν κάποιες ε, ε βασικές υποτυπώδεις ε, υπηρεσίες υγείας στους πληθυσμούς τους. Αυτό, αυτό ζητάμε όταν μιλάμε για ισότητα. Θέλουμε να υπάρχουν περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι, περισσότεροι ε, καταρτισμένοι ιατροί. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στον τον αριθμό των γιατρών, των τεχνικών, των νοσοκόμων που μπορούν να ε, ανταποκριθούν στι ανάγκε του πληθυσμού. Σε σχέση με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει ο ΠΟΗ, έτσι, και πολλά από αυτά συνδέονται με τι επενδύσει. Επενδύσεις ε, ε, σε εσωτερικό επίπεδο αλλά και η μόχλευση διεθνών, διεθνής χρηματοδότησης. Θα κλείσω λέγοντας ότι στον ΠΟΗ, στην περιοχή της Αφρικής, υπάρχει μια ατζέντα για την ε, μεταρρύθμιση, για την αλλαγή. Είναι ένας τρόπος συνεργασίας με τις 47 χώρες της Αφρικής, έτσι ώστε να προσανατολίσουμε καλύτερα τους πόρους μας ε, στις προτεραιότητες που αφορούν την κάθε χώρα, Υπάρχουν χώρε όπω στην Ιγυρία, η Αιθιοπία, η Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και πολύ μικρέ χώρε, όπω το Λεσότο ή στο Σάουτο και Πρίνσιπε, όπου ε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε ε, αυτά που προσφέρουμε στι ανάγκε ε, Στο πρόγραμμα αυτό λοιπόν προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εστίασή μα στο αποτέλεσμα, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην χρήση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μα Και αρχίζουμε να βλέπουμε ε, βελτίωση. Θα ήθελα τελειώντα να πω ότι μαθαίνουμε πολλά από κοινού με τα κράτη-μέλη ε, για το πώς μπορούμε να θεσπίσουμε προγράμματα, ε, συστήματα υγείας που να φέρουν αποτέλεσμα απέναντι στα προβλήματα αυτά. Το να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υπάρχει ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εργαστήκαμε γύρω από το θέμα του διαλόγου ε, στον τομέα της υγείας, στην σωστή διακυβέρνηση στον τομέα αυτών. Είναι πολύ σωστό να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση να αντιμετωπίσουμε τα, ε, τις προτεραιότητες, ε, τα πιο μεγάλα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Υπάρχει και ένα, μια συζήτηση, ένα πρόγραμμα σκέψης, ε, σε ό,τι αφορά την καθολική ιατρική περίθαλψη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for your Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επισκόπηση των προβλημάτων και της καταστάσεως. Οι συνάδελφοι θέλουν να λάβουν το λόγο, θέλουν να σχολιάσουν. Έχουν κάποια ερώτηση, μήπως. Κύριε Τσάλτος. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευρωβουλευτής από την Ιρλανδία. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τι θα κάναμε χωρίς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που θεωρείται δεδομένος όπως και άλλοι φορείς που εργάζονται σε πολλούς τομείς ε, χωρίς να προβάλλονται ιδιαίτερα και τους θεωρούμε στα δεδομένους φορείς, αλλά δεν ξέρω θα κάναμε χωρίς αυτούς. Ερώτηση. Σε ποιο τομέα χρειάζεστε περισσότερους πόρους στη δουλειά που κάνετε στην Αφρική. Απάντηση κυρία Σμαέτη. Ευχαριστώ που μας θυμήσατε ότι πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο τη δουλειά μας χρειαζόμαστε στις χώρες ε, μεγαλύτερο δυναμικό για το έργο του ΠΟΗ. Σε πολλές χώρες έχουμε μικρές ομάδες, λίγους εμπειρογνώμονες. Στα γραφεία μας έχουμε εθνικούς εμπειρογνώμονες που εργάζονται διάφορους τομείς των προγραμμάτων. Θέλουμε να έχουμε υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας στη διαμόρφωση πολιτικής για να συντονίζονται οι προσπάθειες και να βοηθούμε και την κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις να κατευθύνει τις προσπάθειες. Να έχουμε ένα πλαίσιο ούτως ώστε τότε να χορηγηθεί τεχνική υποστήριξη. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δυναμικό σε υψηλό επίπεδο, περισσότερους ανθρώπους με, υψηλές, με γνώση υψηλού επίπεδου. Έχουμε ανθρώπους που είναι ειδικευμένοι σε διάφορους τομείς για τη φυματίωση, για το AIDS, για την ολονοσία. Όλα αυτά πρέπει να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο ενός ευρύθμως λειτουργούντος συστήματος υγείας και πρέπει αυτές οι δυνατότητες να αυξηθούν σε επίπεδο των διαφόρων χωρών. Ευχαριστώ, κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρία μου. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Αγαπητοί συνάδελφος, σαν αδελφοί μας, ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είπατε και το θεμελιώδες που τονίσατε, ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε διαθρωμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, ένα στέρεο σύστημα. Ελήψη αυτού, κάθε προσπάθεια, όσο και αξιέπαινη και αν είναι, δεν θα δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Προφανώς, μπορείτε να μας πείτε αν έχει την καλοσύνη, σε ποιο βαθμό και πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, ούτω ώστε να επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι στόχοι που βασίζονται στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Έτσι θα μπορούμε να προστατεύσουμε όλους τους κατοίκους της Αφρικανικής Υπήρου και θα αποφύγουμε το ξερίζωμα των πληθυσμών, που είναι η μόνη λύση για κάποιου πληθυσμούς, που δεν μπορούν να έχουν περίθαλψη ούτε να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα της υγείας ή διατροφή. Έχουμε κάθε σεβασμό για την Αφρική, μεγάλο σεβασμό και για τους κατοίκους αυτής. Και γι' αυτό σκεφτόμαστε αυτή τη δυνατότητα οι άνθρωποι να μείνουν στη χώρα τους, ε, στις περιοχές τους και στο, στις πολιτισμικές τους παραδόσεις. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω γαλλικά. Όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια και προστασία, πρέπει να γίνουν πολλά για να επηρεαστούν οι διάφοροι πολιτικοί των χωρών και η διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Σαν ΠΟΗ έχουμε εργαλεία και ιδέες για τις τεχνικές πτυχές της εργασίας μας. Πολιτική απόφαση πρωτίστως απαιτείται για να δημιουργηθεί μηχανισμός, μια πλατφόρμα, μια βάση για κοινωνική πρόνοια, για προστασία, να συναθρίζει τις συνεισφορές και των φτωχών και εκείνων που είναι λίγο πιο πλούσιοι και να έχουμε σύστημα που λειτουργεί τον πληθυσμό. Αυτή είναι πολιτική απόφαση και στρατηγική θα έλεγα που κινείται προς την κοινωνική ισότητα. Είναι μια δεντολογική απόφαση. Πρέπει να συνεργαστούμε εμείς με τα εργαλεία μας, με τις κατευθύνσεις που έχουμε. Κάνουν κάποιες δοκιμές στη Ρουάντα, το Μπουρούντι, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Μπορούμε να ακολουθήσουμε και κάποια παραδείγματα και κάποιες εμπειρίες αφρικανικές που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας απευθύνουμε εκκλήσεις από πλευράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και εσείς απευθύνετε εκκλήσεις. Και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στις χώρες αυτές που απευθύνουν εκκλήσεις όσον αφορά τη σωστή χρηματοδότηση της υγείας. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στις κατάλληλες αποφάσεις. Να προστατεύεται ο πληθυσμός και να καταλήξουμε σε κάποια ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση του λαού στις ε, υπηρεσίες περίθαλψης υγείας. Πρέπει να σεβόμαστε πάντα το πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε στις διάφορες χώρες. Τι πιστεύει ο κόσμος πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Μπορούμε να λέμε πολλά στον κόσμο, στο λαό, αν δεν πείθονται όμως. Πώς να το πω. Αν δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που ζουν και με τις πεπιθήσεις τους, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει να τονίσουμε πολύ περισσότερο το διάλογο με τις κοινότητες. Να ακούσουμε τι λέγουν, τι σκέφτονται. Και πρέπει να προσαρμόζουμε τις στρατηγικές μας δεόντως. και να λαμβάνουμε αποφάσεις για την υγεία των πληθυσμών αφού ακούσουμε τις απόψεις τους και τους καταλάβουμε. Από την απάντηση στην επιδημία της έμπολα ε, βρήκαμε κάποιες προσεγγίσεις. Έπρεπε να προσαρμοστούμε στις πρακτικές των κοινοτήτων, να συνεργαστούμε μαζί τους για να εφαρμόσουμε δράσεις που οδηγούν στην, στον έλεγχο αυτής της ασθενείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αναφέρατε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε είναι η έλλειψη γιατρών όσον αφορά την περίθαλψη των ασθενών. Αναφέρατε λοιπόν την έλλειψη των γιατρών, ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, σημαντικότατο πρόβλημα για τη θεραπεία των ασθενών. Και είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που υποχρεώνεστε να επιτρέψετε σε νοσηλεύτριες να αναλάβουν κάποιες ευθύνες που διαφορετικά θα έπρεπε να αναλαμβάνουν μόνο οι γιατροί. Τι είδους λύσεις διαβλέπετε για αυτό το πρόβλημα. Πιστεύετε ότι θα πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά ε, όργανα και οι θεσμοί γενικά θα πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση ε, προσωπικού στην Αφρική. Ε, μήπως μπορούν να διατεθούν πόροι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτως ώστε να εκπαιδεύουν προσωπικό από την Αφρική ή μάλλον ανθρώπους που έρχονται να σπουδάσουν στην Ευρώπη, να γίνονται γιατροί και να επιστρέφουν στην Αφρική και να μπορούν να βοηθάν ε, τον κόσμο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Τι συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ένα ολόκληρο φάσμα λύσεων όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το πρόβλημα που αφορά τους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Συστήναμε ότι πρέπει οι χώρες να αυξήσουν την εκπαίδευση των γιατρών, την κατάρτιση των γιατρών, εντός της χώρας, αλλά και εκτός, στο εξωτερικό, διεθνώς. Παρατηρούμε ότι πολύ συχνά όταν οι εκπαιδευόμενοι αποστέλλονται στο εξωτερικό λόγω των συνθήκων εργασία που επικρατούν στη χώρα καταγωγής δεν επιστρέφουν. Μένουν στη χώρα στην οποία πήγαν να εκπαιδευτούν. Αλλά οι χώρες ε, πρέπει να αυξήσουν ε, τις δυνατότητε κατάρτιση. Υπάρχουν και ε, κενά όσον αφορά τους γιατρούς. Δεν αρκεί η εκπαίδευση. Αυτοί οι γιατροί πρέπει να απορροφούνται όμως, να απορροφούνται στο σύστημα. Να απασχολούνται. Αυτό εξαρτάται πολύ από, τα, από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και το δημόσιο τομέα, τη δίκηση και τα όρια που έχουν, πόροι, θέσεις που είναι διαθέσιμες στις χώρες. Αυτά είναι προβλήματα. Έχουμε ένα πρόγραμμα υποστήριξη για να στηρίξουμε τις χώρες να επανεξετάσουν το φάσμα των δράσεων, να δουν πώς μπορούν να βελτιώσουν και την κατάρτιση και την συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες, ούτως ώστε να βελτιωθεί μειωθεί ο αριθμός του προσωπικού και οι συνθήκες εργασίας. Διότι έτσι ε, θα, μπορούμε να, θα μπορούν οι χώρες να κρατήσουν κόσμο στις χώρες. Έχουμε πρόβλημα κατανομής των γιατρών στις ε, χώρες της Αφρικής. Έχουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου. Τη δουλειά των γιατρών στην Ήπεθρο την αναλαμβάνουν περισσότερο οι νοσοκόμες, γιατί υπάρχουν ελάχιστοι γιατροί. Ε, πρέπει να εκπαιδεύσουμε και παραϊατρικό προσωπικό. Όσο γίνεται η προσπάθεια αυξήσεως του αριθμού των γιατρών. Χρειάζεται και πιο άμεση δράση για να καλυφθούν τα κενά όσον αφορά τη δυνατότητα παροχής ε, βασικών ε, υπηρεσιών υγείας του πληθυσμού. Και πρέπει και άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού να βοηθούν τους γιατρούς και να λαμβάνονται τα καθήκοντα. Υπάρχει ε, μία ανακατάταξη καθηκόντων. Χρειάζεται σωστή επιτήρηση. Με σωστή επιτήρηση μπορεί, παραδείγματος χάρη το AIDS, να δώσει σωστή κάλυψη. Προσωπικό ε, ιατρικών επαγγελμάτων να πραγματοποιεί και σε τομέ και λοιπά στην Ήπεθρο και σε περιοχέ που έχουν ελλείψει γιατρών. Μπορούν να καλυφθούν τα κενά. Ε, γνωρίζετε ότι χρειάζεται επαφή με τι κοινότητε. να γίνεται πρόληψη, πρόθεση, ενημέρωση από μέλη της κοινότητας. Στα σπίτια, στα νοικοκυριά μπορεί να γίνει, σε επίπεδο κοινότητας. Πρέπει να εκπαιδεύουμε τον κόσμο επιτόπου. Θέλουμε μεν να φτάσουμε στα πρότυπα του ΠΟΕ για τους γιατρούς, για τις ΜΕΣ, για τους νοσηλευτές. Παράλληλα όμως συστήνουμε κάποιες στρατηγικές για να καλύψουμε κατεπίγουσες ανάγκες για κατάρτιση, εποπτεία, για να εκτελούν οι άνθρωποι κάποια καθήκοντα, ούτως ώστε να αυξάνεται το τρόπος η δυνατότητα να περιθάλπουμε κόσμο. Ε, πρέπει βέβαια να προωθούμε και την καριέρα των ε, μελών των παραγιατρικών επαγγελμάτων που μπορούν να εκτελούν διάφορα καθήκοντα όπως οι κυσαρικές τομές κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούμε λοιπόν αυτά που μας λέτε. Αμάλλον ακούμε στις ειδήσει ότι σημειώνονται, έχουμε έκρηξη νέων πολέμων στην Αφρική δυστυχώς. Υπάρχουν χώρες όπου οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να διατηρήσουν καν τη σταθερότητα, να λειτουργήσουν σταθερά. Υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των φυλών ή ανατρέπονται τα καθεστώτα, κυβερνήσεις. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε, τι δυνατότητες υπάρχουν. Υπάρχουν δυνατότητες για να εκτελούνται οι αποστολές αυτές περίθαλψης που αναφέρατε όταν υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα και αυτή η αστάθεια. Αν κυρία Μαέτη απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όταν η κυβέρνηση έχει προβλήματα όσον αφορά την οργάνωση να επιβληθεί, όταν υπάρχουν συγκρούσεις, εξεγέρσεις, Υπάρχουν πολλές χώρες που συμβαίνει αυτό επί παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Και βλέπουμε ότι η διεθνής κοινότητα και οι συνεργαζόμενες κυβερνήσεις και οι διεθνείς φορείς και οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών προσπαθούν να βοηθήσουν για την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και αυτό που κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σαν φορέας είναι να συντονίζουμε το έργο των διαφόρων που συμμετέχουν στον τομέα της υγείας εκπαίδευση, νερό, υγεία κλπ. για να παρασχεθούν οι βασικές υπηρεσίες στον πληθυσμό και να μείνει ο κόσμος ζωντανός. Τα παιδιά να εκπαιδεύονται. Ο ρόλος που παίζουμε συνεργαζόμενοι μάλλον σε του του ΟΗΕ και της κυβέρνησης ποιος είναι. Προσπαθούμε να συντονίσουμε τις διάφορες συνεισφορές όλων αυτών των φορέων με έναν τρόπο που να υπάρχει εξορθολογισμένη αντιμετώπιση της ανάγκης του πληθυσμού για την υγεία, για τους εμβολιασμού κλπ. και την αντιμετώπιση ε, διαφόρων ε, νόσων. Αυτό κάνει ο ΠΟΗ σαν τεχνικός φορέας. Σε αυτές τις περιστάσεις κινούμεθα υπό την αιγίδα ενό συντονιστού του ΟΗΕ για να αντιμετωπίσουμε περίπλοκες κατεπίγουσες ανάγκες και εμεί εκεί εντασσόμεθα σε αυτό το πλαίσιο. Προσπαθούμε να ηγηθούμε και να συντονίσουμε το έργο του τομέα Υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωποι του Αφρικανικού Κοινοβουλίου έχουν το λόγο τώρα. Ο κ. Τουρίας Κάλι από το Κοινοβούλιο του Μαρόκου έχει το λόγο. Ε, δεν σας βλέπω που βρισκόσαστε. Κυρία. Η κυρία Κάλλη. Κυρία Πρόεδρα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που καλέσατε την αντιπροσωπεία του Μαρόκου για να συμμετάσχει στην ανταλλαγή απόψεων στον αφορά ε, τις μεταδοτικές ασθένειες. Όπως υπογράμμισε η κυρία Μωέτη, σημασία έχει καταπολέμηση της τη, ε, της μητρικής διότι η υγεία των γυναικών αντιπροσωπεύει και τη θέση της γυναίκας σε συγκεκριμένη κοινωνία στο Μαρόκο. Κάναμε συνεχώς προσπάθειες και αυτές επέτρεψαν τη μείωση του ποσοστού από 35% κατά 35% την τελευταία πενταετία της νησιμότητας των γυναικών, των μητέρων. Είναι ψηλό το ποσοστό, 112 θάνατοι στις 100.000 μητέρες. Μειώθηκε όμως σύμφωνα με την τελευταία έρευνα κατά 72%. Μια άλλη πτυχή που υπογράμμισε κάποιος ευρωβουλευτής είναι η ιατρική περίθαλψη. Η κάλυψη η ιατρική αυξάνεται σημαντικά πλευράς νομοθετική στη χώρα μας 90% του πληθυσμού θα έχει δικαίωμα σε μια κάλυψη ιατρική και σύνταξη και κοινωνική σφορά ε, η συνεισφορά επιτρέπει να προστατεύονται από την ε, περιθωριοποίηση και τη μη κάλυψη των τομέα υγείας. 6,5% ε, ε, είναι πολύ χαλημένο το ποσοστό. Ε, δεν δίνουμε πολλά χρήματα ενισότητα όσον αφορά την περίθαλψη, κυρίως στην Ήπεθρο. Παρ' όλα αυτά, το Μαρόκο διαθέτει προγράμματα στον τομέα της προστασίας της υγείας και του ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών και των αδειωμένων ασθενειών για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να συμβάλλει και στις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα αυτό. Αυτές οι προσπάθειες που υπογραμμίζονται από τον ΠΟΗ, κυρίως στην αντιμετώπιση της επιδημίας της έμπολα κατεβλήθησαν. Οι μεταδοτικές ασθένειες ε, είναι θέμα δημόσιας υγείας στο Μαρόκο. Συνδέονται συνήθως ασθένειες με τη φτώχεια και με τους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως των μεταναστών, που γίνονται δεκτοί και που εντάσσονται στο Μαρόκο και τους προστατεύουμε, τους καλύπτουμε. Όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες έχουμε τις περιπτώσεις που καλύπτουμε. Εκεί όπου η ασθένεια μεταδοτική ελέγχεται και θεραπεύεται, όπως η λονοσία, σχιστοστομία, χόλερα, η ε, επιπεφική της των νεογνών και κάποιες ασθένειες που μπορούν να αποτελέσουν το εμβολιασμού. Ο εμβολιασμό είναι πάρα πολύ επιτυχής. 95% έχουμε κάλυψη μέσω των εμβολιασμών. Δεύτερη κατηγορία τώρα που καταβάλλονται προσπάθειες και παρά τις προσπάθειες ε, υπάρχει μετάδοση των ασθενειών, είναι η φυματίωση, ε, μηνυγκίτιδε, λησμανίωση που επανέρχεται, διάφορα προβλήματα του ανθρωπιστικού συστήματος, διατροφικές ε, δηλητηριάσει, υπατήτηδα τρίτη κατηγορία. Έχουμε αναδυόμενα προβλήματα της υγείας, όπου εκεί τα μέτρα είναι ανεπαρκή ή που ξαναεμφανίζονται προβλήματα. Λοιπόν, η φυματίωση είναι ένα πρόβλημα που επιμένει, σημαντικό πρόβλημα η δημόσια υγεία. 27 με 28.000 νέα κρούσματα το χρόνο, κυρίως της πόλης και 200 περίπου κρούσματα που ε, αντιστέκονται αυτές οι περιπτώσεις ε, στα αντιβιωτικά και η λησμανίωση επίσης είναι πρόβλημα, κυρίως στα αστικά κέντρα, ε, υψηλός αριθμός των κρούσματων. Πάνω από 6.500 περιπτώσεις. Η μηνυγκίτιδα επίσης ε, σποραδικά εμφανίζεται οδηγεί σε υψηλό αριθμό θανάτων, περίπου 8 με 12% από τα κρούσματα και άλλε ασθένειε. Λεπτοσπύρωση, παραδείγματο χάρη, είναι πρόβλημα. Παρακολουθείτε επιδημιολογικά συνεχώς. Δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται. Αυτές που ελέγχονται, εξαλείφονται όπω η χιστοστομίαση, η επιπεφική της, το τράχωμα, ε, ε εντάσσονται σε στρατηγική ε, συντήρηση καταστάσεως ε, το AIDS τώρα. Σε εθνικό επίπεδο έχουμε στρατηγική. Έχουμε συνοδευτικό σχέδιο. Το 86 με τελευταίο ασθενή. Μετά είχαμε 6.000 περιπτώσεις που διαγνώστηκαν το 2010. 50% ήταν οι γυναίκες. Μετάδοση κυρίως ε, από σεξουαλικές σχέσεις ε, και από ναρκωτικά. Έγιναν σοβαρές προσπάθειες. Εκστρατείες πρόληψης στις γυναίκες και στους νέους. Ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ευάλωτες ομάδες. Πρόσβαση στην πρόληψη ε, για τη μετάδοση από μητέρα στα παιδιά και μέτρα για την ε, τυχαία έκθεση ή μέσω σεξουαλικής επαφής στον ιό του AIDS στα νοσοκομεία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τη θεραπεία των ατόμων που είναι φορείς αλλά καλύπτουμε το 48% των ασθενών το 2016 καλύψαμε έναντι 16% το 2010. Είχαμε κάποια πρόοδο, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια. Υπάρχει εθνικό πρόγραμμα ψυχολογικής και κοινωνικής ε, συνοδείας και υποστήριξης μαζί με τα κοινοτικά συστήματα που υπάρχουν για να διευκολύνουμε την δράση των ΜΚΟ στους τομείς. Όλα αυτά για να πετύχουμε το γενικό στόχο του ΟΗΕ για το AIDS, δηλαδή μια μείωση κατά 75% από τώρα μέχρι το 2020 σημαντική τροχοπέδη για την επίτευξη του στόχου είναι ο στιγματισμός και η ποινικοποίηση ε, των ανθρώπων που πάσχουν από αυτό και είναι η μελανή κοιλίδα. Είναι βάρωτοι πληθυσμοί που αντιπροσωπεύουν το 80% των ε, ασθενών, άντρες, ομοφιλόφιλους, ε, πόρνες, μετανάστες κλπ. Αυτή είναι η σφαιρική γενική εικόνα όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες. Ε, συνεργαζόμαστε ε, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για να αξιολογήσουμε μαζί με το Υπουργείο το αρμόδιο ε, την προστασία της δημόσιας υγείας, να βελτιώσουμε την απόδοση των διαφόρων πολιτικών που ασκούμε για την προστασία της υγείας και να αναπτύξουμε ένα, μια στρατηγική για τον έλεγχο της υγείας και που είναι, θα είναι δυσυνοριακός. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ρουσιαστή Αλή Ουαϊκίκη από την Κοινοβουλευτική Σύνοψη της Νιγηρίας. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει ε, ένα ρητό στην Αφρική ε, και στην Ιγυρία που λέει ότι η υγεία είναι πλούτος. Και εμείς λοιπόν στη δική μου χώρα στην Ιγυρία έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να βελτιώσουμε την κατάσταση υγείας των, ανθρώπων, των, των πολιτών μας μέσω καλύτερων υγειονομικών συνθήκων, μέσω πρόσβασης σε πόσιμο νερό, μέσα, ε, μέσω πρόσβασης σε βασικές ε, υποδομές ε, νοσοκομιακές και σε βασική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και εμείς ως κυβέρνηση και ως κοινοβούλιο, ως κοινοβουλευτική συνέλευση, έχουμε θεσπίσει ένα νόμο στον οποίο προβλέπεται ότι ένα, το 1% των όλων των εσόδων που εξέρχονται στην Ιγυρία ε, κατευθύνεται προς ένα ενοποιημένο ταμείο ε, το οποίο μοιράζονται διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες αλλά ε, μέσω του οποίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις για φαρμακευτικέ ε, υπηρεσίε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μοέτη για τα στατιστικά στοιχεία που μας παρουσίασε, αλλά ε, ε, δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται βέβαια σε αυτές τις κατάξεις εδώ η κυρία. Πάντως εμείς έχουμε θεσπίσει ένα σχετικό νόμο για τη δημιουργία αυτού του ενοποιημένου ασφαλιστικού ταμείου, όπου έχουμε ε, ε, τη συμμετοχή τη ομοσπονδιακή κυβέρνηση και 48 περιφερειακέ κυβερνήσει που συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο και όπου ε, οι προτεραιότητες αυτές σε ό,τι αφορά το ταμείο μοιράζονται τόσο από πλευρά των περιφερειακών κυβερνήσεων όσο και από πλευρά της κοινοβουλευτική συνάδευσης. Μέσω λοιπόν αυτού του, κοινο, του ενοποιημένου δηλαδή ασφαλιστικού ταμείου έχουμε δημιουργήσει και ένα πρόγραμμα για τον, ε, για τον έλεγχο ε, του AIDS στην Ιγυρία. Ε, και βέβαια κάποιοι από εσά, από του εταίρου μα δηλαδή και από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είχατε επαφή με αυτόν τον φορέα, προκειμένου δηλαδή ε, να καταπολεμήσουμε τις, τον αντίκτυπο τη επιπτώσει του AIDS. και έχουμε πραγματικά οδηγηθεί σε επιτυχίε. και επίση έχουμε μέσω της Ένωσης της Νιγηρίας δημιουργήσει κάποιες ε, ε, νοσοκομικές υποδομές που παρέχουν ποιοτικέ υπηρεσίες στους πολίτες μας αλλά και ανθρώπινο ε, και εκπαίδευση στο ιατρικό και παραγωγικό προσωπικό. Και οι δύο βασικέ θετικέ οργανώσει στην Νιγηρία είμαστε τυχεροί για το γεγονό ότι έχουν δημιουργήσει και έχουν συμβάλει στην δημιουργία ε, κάποιων ε, μορφωτικών ιδρυμάτων, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, εκπαίδευση ακριβώς τέτοιου παραγωγικού προσωπικού, αλλά για παράδειγμα από το τομέα των οδοντιατρικών, γενικά το τομέα της φροντίδας και ούτω καθεξής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ελονοσία, η οποία σήμερα είναι πιο θανατηφόρα από ότι το AIDS, έχουμε ξεκινήσει εδώ προσπάθειες, για παράδειγμα, μέσω της παροχής αποστηρωμένων έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση τη υγεία των πολιτών μα όπου και αν αυτοί διαμένουν. Και να, ε, δηλαδή, λάβουμε προληπτικού χαρακτήρα δράση. Και επίση, ω Κοινοβούλιο, έχουμε θεσπίσει μια νομοθεσία όπου ε, τα απαραίτητα φάρμακα, η απαραίτητη περίθαλψη μπορεί να δίνεται σε ε, άτομα με αναπηρία και σε άλλα ευάλωτα άτομα, όπως επίσης και παροχή σε μέσα μεταφορής και ούτω καθεξής. Επίσης έχουμε δημιουργήσει και μια υπηρεσία σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ακριβώς αφορά στην πρωτοβάθμια αντιμετώπιση, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη των ε, πολιτών. Και προβλέπεται ότι από το 2019 όλοι οι νοσοκομιακοί δηλαδή 25.000 στην Νιγηρία, θα περιλαμβάνουν εφεξή και ακριβώς ένα ε, τομέα, ένα κέντρο πρωτοβάθμιας ε, περιθαλψής. Και επίσης υπάρχει και ένα ε, ταμείο παρέμβασης μέσω του οποίου δεν θα υπάρχει ο ανταγωνισμό πλέον μεταξύ των περιφερειακών οργανώσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτή την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Με τη δημιουργία δηλαδή των κέντρων σε όλου του νοσοκομιακού ε, θαλάμου, θα υπάρχει αυτή η πρωτοβάθμια περίθαλψη σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα νοσοκομεία. Από εκεί και μετά έχουμε μια νέα προσέγγιση η οποία ε, προστοχεύει στην αντιμετώπιση τη ε, ανεργία των νέων ειδικότερα και προκειμένου ε, ε, εκείνοι οι τελειόφοιτοι για παράδειγμα, οι οποίοι όμως δεν έχουν κάποια δουλειά, μπορούν για παράδειγμα να συμπληρώσουν μια ε, εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορούν να εργαστούν για παράδειγμα ως εργαζόμενοι στις κοινότητες, ως παραδοτικό προσωπικό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της μη απασχόλησης ταυτόχρονα με το πρόβλημα της εκμάθησης μιας πιο υγιεινής ζωής. Πώς να δηλαδή ζει κανείς μια πιο υγιεινή ζωή. Επίσης, ο νέος πρόεδρος της κυβέρνησής μας ε, φρόντισε κάθε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να λάβει 1,5 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια ούτως ώστε να ε, επενδύσει στους, στις, ε, στους φορείς της υγείας. Και ο Γενικός Γραμματέας Τη παγκόσμια Οργάνωση υγεία ε, είχε ε, εμπιστευτεί την Ιγερία και είχε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Και αναφέρθηκε και το ζήτημα της συνεργασίας όχι μόνο σε ό,τι αφορά το AIDS, για παράδειγμα, ε, αναφερθήκαμε γενικότερα στα ζητήματα της κοινή ενίσχυσης ε, των δομών μας, ε, των ε, δικτύων συνεργασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να βρεθούμε στην ίδια κατάσταση σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας που βρίσκονται οι πιο ανεπτυγμένες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ναι, να δώσω λέω πρόεδρος το λόγο στην δόκτωρα Μοέτη σε περίπτωση που θέλει να σχολιάσει ε, κάποια από τα στοιχεία που υπόθηκαν από την πλευρά των συναδέλφων από τα κοινοβουλία της Αφρικής. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω του προσώπους των κοινοβουλίων του Μάρκου και τη Αφρική ε, για τα όσα μοιράστηκαν μαζί μα προ τα όσα έχουν κάνει προκειμένου να παράσχουν η περιθάλψη στου πολίτε του ε, και που αναφέρθηκαν στι επιτυχίε και στα προγράμματα που έχουν λάβει η χώρα στο Μαρόκο και στην Ιγυρία. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη μετρική τη νημότητα, αλλά και τα όσα αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην ε, Ιγυρία για την αναβίωση, αν θέλετε, του σε της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ε, από τότε που ε, έγινα περιφερειακή διευθύντρια, ε, έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές στην Ιγυρία, μάλλον περισσότερο από κάθε άλλη χώρα και βρέθηκα και πάλι πρόσφατα εκεί στο πλαίσιο μια κατά της πολιομελίτιδας και της ελονοσίας αλλά και σε ό,τι αφορά την επαναδημιουργία, την ανασύσταση κάποιων δομών ε, υγείας ε, εκεί. Οπότε ε, συνεργαζόμαστε εντατικά και με το Υπουργείο Υγεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο αλλά και με του διαφόρους κυβερνήτε σε περιφερειακό επίπεδο ακριβώ για την περίθαλψη τη πρωτοβάθμια πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την αναζωογόνηση αυτού του τομέα καθώ και άλλα σχετικά προγράμματα όπω αυτό τη καταπολέμηση τη ελληνονοσίας και σε σχέση με μια σειρά από περαιτέρω ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε. Νομίζω πω η στρατηγική στην οποία αναφερθήκατε για την αξιοποίηση δηλαδή του δυναμικού των νέων και το πώς αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν στον ε, τομέα ακριβώ τη υγεία είναι πραγματικά μια πολύ εύστοχη προσέγγιση. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει και στην ενίσχυση του τομέα τη υγεία σε αυτέ τι χώρε και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι και εμεί ε, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση των διαβόλων ε, δομών, των θεσμικών δομών στην Ιγυρία προκειμένου να καταστεί δυνατή η βελτίωση αυτή δηλαδή της ποιότητας του του επίπεδου εκπαίδευση του ε, προσωπικού στον τομέα τη υγεία, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλουν καλύτερα και στην, στο να σώνουν ζωέ τελικά. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκλησή σα ε, σήμερα εδώ για να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα και, να, και αυτά τα σχόλια και να σα πω ότι στο πλαίσιο τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, Αφρικανική Ένωση, ειδικότερα δε στο επίπεδο των ε, βουλευτών, το ζήτημα ειδικότερα της απαραίτητης χρηματοδότηση και του κατάλληλου κατάλληλου τύπου χρηματοδότησης, για παράδειγμα μείωση δηλαδή του οικονομικού άχθους για την πρόσβαση στην πρωτοβάθμια ε, περίθαλψη, αλλά και για παράδειγμα την ε, πολυδιάστατη εδώ προσπάθεια σε μια σειρά από αναπτυσσόμενους ε, τομείς ανάπτυξης μάλλον είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει κατάλληλη ε, συνεργασία ανάμεσα στους διαφορούς τομείς έτσι ώστε να άλλο υποστηρίζονται και κάτι τέτοιο βέβαια είναι ιδιαίτερα χρήσιμο έτσι ώστε και εσείς να βοηθάτε την εκτελεστική αν θέλετε εξουσία να λαμβάνει τις σωστές ε, αποφάσεις ε, και να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Δηλαδή αυτό το κάνετε ήδη αλλά και αυτό ζητούμε και εμείς από τη δική μας πλευρά. Ως τεχνική δηλαδή υπηρεσία βρισκόμαστε ω Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία στη διάθεσή σα για να παρέχουμε ε, έμπειρο γνωμοσύνη, στοιχεία και τι πληροφορίε ε, που, ε, που χρειάζονται τα κοινοβούλια έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ του και έτσι να σώμουν περισσότερε ανθρώπινε ζωέ. Σα ευχαριστούμε πολύ, Δ. Μοέτη. Και βέβαια, όποτε θα έχετε και πάλι κάποιε εργασίε εδώ στι Βρυξέλλε, θα σα καλέσουμε και πάλι για να μα πείτε πώ εξελίσσονται οι εργασίε σα. Και βέβαια σα ε, βεβαιώνουμε ότι έχετε την αμέριστη υποστήριξη μα. Σα ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Συνάδελφοι, τώρα θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σε ό,τι αφορά ε, το πακέτο για τις ε, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες ε, οδήγησης. Το τέταρτο λοιπόν πακέτο για αυτές τις εκπομπές ε, συζητείται αυτή την περίοδο στην τεχνική ομάδα εργασίας για τις ε, εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για τα ελαφρά οχήματα και προβλέπει μια σειρά από τεστ σε ό,τι αφορά ακριβώ την χρήση τέτοιου είδου δοκιμών και το πώ μπορούν να επιτευχθούν μερόληπτε ανεξάρτητε δοκιμέ. Επίση, συζητούνται μια σειρά από ζητήματα που είχαν παραμείνει σε εκκρεμότητα στο πλαίσιο των τριών περασμένων πακέτων. Από την πλευρά λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουμε κάποιους την, κυρία Σικόφκα από την ε, Γενική Διεύθυνση Grow και τη μονάδα σε ό,τι αφορά ακριβώς ε, των εκπομπών των, από τα αυτοκίνητα. Της δίνουμε λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις εργασίες που έχουμε κάνει έως τώρα σε ό,τι αφορά το τέταρτο πακέτο για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και να σας δώσω μια γενική πληροφορία εδώ, ένα γενικό υπόβαθρο. Ίσως θα θυμόσαστε ότι τον περασμένο Μάιο οι δοκιμές σε ό,τι αφορά τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης έχουν αρχίσει να ισχύουν από το Σεπτέμβριο πλέον σε, τα, σε ό,τι αφορά τους νέους τύπους οχημάτων και από εκεί και μετά στο ενδιάμεσο διάστημα έχουμε στο τρίτο πακέτο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των σωματιδίων και αυτή την περίοδο οριστικοποιούμε τι εργασίες μα σε ό,τι αφορά τι πραγματικέ συνθήκε οδήγηση, σε ό,τι αφορά δηλαδή, τη συμμόρφωση των σχετικών δοκιμών. Θα θέλαμε τώρα να σα ενημερώσουμε σε ό,τι αφορά το τι κάνουμε αυτή την περίοδο και σα ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία. Είχαμε κάνει δηλαδή έναν διάλογο πέρυσι στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου και τον είχαμε βρει πολύ χρήσιμο. Οπότε στο ίδιο πνεύμα θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση σήμερα σε ό,τι αφορά το τέταρτο πακέτο. Υπάρχουν μία σειρά από ζητήματα τα οποία θα καλύψουμε στην νομοθεσία που επικοιτά και εδώ βλέπετε στη διαφάνεια τα κυριότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Καταρχήν λοιπόν θα εξετάσουμε το πώς να επαληθεύουμε ε, την χρήση των αυτοκινήτων, δηλαδή αυτό το in-service conformity όπως το βλέπετε, δηλαδή κανόνες που θα ε, διασφαλίζουν ότι τα αυτοκίνητα ε, συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα με βάση τα οποία έχουν εγκριθεί. Και επίσης θα υπάρξουν νέες ε, ε, μέθοδοι ε, αξιοποίησης ό,τι αφορά τις εκπομπές και επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και κάτι καινούριο, το περιθώριο, το margin. Είχαμε προβλέψει στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου, αν θυμόσαστε, ένα προσωρινό περιθώριο, η conformity factor όπως λεγόταν, παράγοντας συμμόρφωσης, ε, και μετά ένα δεύτερο ε, περιθώριο και αυτό το δεύτερο περιθώριο είναι όπου θα αναθεωρήσουμε στο πλαίσιο του τέταρτου πακέτου. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό PEMS, δηλαδή αυτόν τον ε, εξοπλισμό για τη μέτρηση των διαφόρων εκπομπών και επίσης θα ασχοληθούμε με κάποια ακόμα ζητήματα με τα οποία δεν είχαμε ασχοληθεί εκτενώς στο πλαίσιο των προηγούμενων πακέτων για παράδειγμα μέθοδοι ε, δοκιμές για τα υβριδικά, βαριακά και το καθεξής. Αυτά λοιπόν εν ολίγης ως προς το τι θα αναθεωρήσουμε στην αρμοθεσία τώρα. Θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το in-service conformity, αυτή η in-service συμμόρφωση. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα θα ε, συμμορφώνονται ε, με τα πρότυπα στο πλαίσιο ολόκληρου του κύκλου ζωής τους, τα πρότυπα αυτά ε, υπό τα οποία έχουν εγκριθεί. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες από όλα τα αισθήματα, PEMS, SEMS, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους εφορεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν θα βασίζομαστε πλέον στις πληροφορίες μόνο από την πλευρά των κατασκευαστών, αλλά και από την πλευρά τρίτων φορέων. Και όταν λέμε τρίτη φορή, μη κυβερνητικέ οργανώσει, οργανώσει των καταναλωτών, περιφέρειε και πόλει, οποιοδήποτε μπορεί να μα παράσχει πληροφορίε. Και θα επαληθεύουμε βέβαια εμεί αυτά τα στοιχεία, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να έχουμε μη αξιόπιστα δεδομένα. Άρα λοιπόν ε, ε, αυτή την περίοδο εξετάζουμε το πώς θα επαληθεύουμε αυτά τα δεδομένα που θα έχουμε συλλέξει και στη συνέχεια θα δημοσιοποιούνται αυτά τα δεδομένα άπαξ ετησίω. Προφανώ θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται περισσότερε φορά, αλλά μία φορά το χρόνο θα ε, δημοσιεύονται. Ε, Τώρα, ε, Καταρχήν, αυτά τα δεδομένα θα ε, αξιοποιούνται για το in-service conformity, αλλά ταυτόχρονα θα αξιοποιούνται και για τις έρευνε σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, κάποιε παρποιήσεις που έγιναν σε ό,τι αφορά του μηχανισμού μετρήσεις, αλλά και Ε, και έρευνε σε ό,τι αφορά τα ε, devices, πάντοτε στο πλαίσιο της ε, εποπτείας της αγοράς, του market surveillance. μία ακόμα διαφάνεια, η οποία δείχνει κάπως περίπλοκη, αλλά δεν είναι τόσο περίπλοκη, μας δείχνει ποιοι θα είναι αρμόδιοι φορείς εδώ. θα έχουμε καταρχήν εκείνους οι οποίοι θα μας απαρέχουν τα σχετικά δεδομένα, όπως είπαμε εδώ θα έχουμε και τρίτους φορείς και από εκεί και μετά μόλις θα επαληθεύονται τα δεδομένα, όπως βλέπετε δηλαδή στο πάνω δεξί ε, κουτί θα υπάρχει η επαλήθευση όπως βλέπετε εδώ στο πράσινο πλαίσιο ε, ε, επαλήθευση δηλαδή στοιχείων σε ό,τι αφορά οικογένειας αυτοκινήτων που θα γίνονται και από ανεξάρτητους ελεγκτέ ή φορεί δοκιμή. Δηλαδή, εδώ και πάλι μπορούμε να έχουμε μία σειρά από διαφορετικού φορεί, έστω και μη κυβερνητικέ οργανώσει, οποιοδήποτε ο οποίο έχει επαληθευτεί όμω και αυτό είναι σημαντικό. Θα χρειάζεται επαλήθευση του ώστε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των σχετικών δεδομένων. Δηλαδή αυτοί οι ανεξάρτητοι ε, φορεί δοκιμή θα πρέπει να έχουν επαληθευτεί. Με βάση λοιπόν αυτέ τι πληροφορίε, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία για μη συμμόρφωση κάποιου οχήματο, θα ξεκινάει μία ε, έρευνα και αν πράγματι αποδειχθεί ότι ένα όχημα δεν συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, ο κατασκευαστής ε, θα οφείλει να προβαίνει σε ε, μέτρα αποκατάστασης αυτής της μη συμμόρφωσης. Και βέβαια η τα αποτελέσματα της έρευνας σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα αυτής της αποκατάστασης θα δημοσιοποιείται. Ε, βέβαια υπάρχουν μια σειρά από ερωτήματα που προσπαθούμε να απαντήσουμε και να επιλύσουμε ε, παρότι βέβαια η βασική μας προσέγγιση είναι αυτή που βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Θα επανέλθω λοιπόν σε αυτήν την ε, δομή στο τέλος της παρουσίασής μου. Το δεύτερο τώρα στοιχείο στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο εξετάζουμε αυτή την περίοδο είναι η καταλληλότητα των μεθόδων ε, αξιολόγησης, ε, δηλαδή το πώς θα αξιολογούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε. Με βάση την εμπειρία μας ε, δεν έχουμε τα κατάλληλα αξιολόγηση αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Δεν είναι δηλαδή εκείνα τα οποία μας παρέχουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Οπότε προσπαθούμε να διερευνήσουμε έναν τρίτο τρόπο, μια τρίτη μέθοδο αξιολόγησης αυτών των δεδομένων. Ε, εξετάζουμε δηλαδή αυτή την περίοδο την δυνατότητα να εξετάζουμε τα αρχικά αυτά δεδομένα, τα raw data, αλλά σε κάθε περίπτωση ε, θέλουμε εδώ να εστιάσουμε στα δεδομένα εκείνα τα οποία ε, δεν είναι ξεκάθαρα και δεν είναι πλήρως αξιόπιστα. Όπως σας είπαμε, θα επιτρέπουμε τώρα και σε τρίτους φορείς να προβαίνουν σε δοκιμές και κατά συνέπεια αυτό χρήζει καθοδήγησης έτσι ώστε δηλαδή όσοι θα προβαίνουν σε τέτοιου είδους δοκιμές σε PEMS θα βοηθάει λοιπόν όσου προβαίνουν σε τέτοιου είδου δοκιμέ, γιατί βέβαια η εμπειρία έχει δείξει ότι υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικέ ε, χρήσει ε, ε, του εξοπλισμού. Οπότε προετοιμάζουμε μια σειρά από εγχειρίδια, ούτω ώστε να υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση και έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι αξιοποιούν ε, αυτά τα πέμψη για τι δοκιμέ, είτε είναι κατασκευαστέ είτε τρίτη φορή να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Και καθώ αναφερόμαστε σε αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να αναφέρω σε κάτι το οποίο είναι ίσω ενδιαφέρον για εσά. Ίσως, ε, ε, θα θυμόσαστε ότι είχαμε υιοθετήσει ε, καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τα, τις συσκευές PIMS και υπήρξε ήδη καθοδήγηση και αυτή την καθοδήγηση προβλέπουμε τώρα να την συμπεριλάβουμε στο τέταρτο πακέτο. και σε ό,τι αφορά τα τη βάση ειδικότερα θα είναι υποχρεωτική η χρήση τους, δηλαδή η καθοδήγηση θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, δεν θα είναι απλώς ε, ε, εθελοντική η χρήση της καθοδήγηση σε ό,τι αφορά τα τη βάση. Κάτι ακόμα, ένα ακόμα στοιχείο που περιλαμβάνεται στο τέταρτο ε, πακέτο είναι η αναθεώρηση, θεώρηση, επανεξέταση αν θέλετε του περιθωρίου. Όπως σας είπα έχουμε δύο περιθώρια σε αυτές τις ε, στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις δοκιμές ε, για τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Έχουμε καταρχήν το πρώτο περιθώριο, το οποίο αφορά την, ε, τις επιδόσεις των ΠΕΜΣ και είμαστε υποχρεωμένοι να, να επανεξετάζουμε ένα πέντε έτη αυτό το περιθώριο. Υπάρχουν μια σειρά από βεβαιότητες τις οποίες προσπαθούμε να εξετάσουμε τώρα, δηλαδή να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι αβεβαιότητε σε ό,τι αφορά τι μετρήσει, ω προ την ε, αξιοπιστία τη μέτρηση των συγκεντρώσεων ε, με βάση την απόσταση του, του μηχανισμού από την πηγή και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά από συντελεστέ εδώ ε, οι οποίοι συμβάλλουν και ο στόχος αυτής της διαφάνειας είναι να σας δείξουμε ότι εξετάζουμε πολύ λεπτομερή τρόπο πώς λειτουργούν τα PEMS και κατά συνέπεια τι μπορεί να έχει επίπτωση στον τρόπο που λειτουργούν και τι αυτό με τη σειρά του μπορεί να έχει επίπτωση στην μέτρηση των εκπομπών. Είχαμε και μια έκθεση που συνέταξε το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το JRC, ε, αρχές ε, Νοεμβρίου και με βάση αυτή την έκθεση θα εξετάσουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να μειώσουμε το σχετικό περιθώριο. Ε, ήδη στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου εμείς καταστήσαμε πιο αυστηρούς τους κανόνες σε ό,τι αφορά τους, ε, τον εξοπλισμό πέμψε, Δηλαδή, ε, έχουμε από τη μία πλευρά κάποια περιθώρια, από την άλλη πλευρά έχουμε και παραμέτρους σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον εξοπλισμό πέμψε και εμείς λοιπόν αρχίσαμε να καθιστούμε και τους κανόνες σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον εξοπλισμό ΠΕΜΣ ε, πιο αυστηρούς. Τώρα, και το τελευταίο στοιχείο για το οποίο θα ήθελα να σα ενημερώσω στο πλαίσιο του τέταρτου πακέτου είναι η εγμόνιση κάποιων προτύπων σε ό,τι αφορά όλα τα POMS, δηλαδή, PEMS. Δηλαδή, θέλουμε όλα τα, όλος ο εξοπλισμός, όλα τα tools σε ό,τι αφορά τα PEMS να ακολουθούν τις ίδιες προδιαγραφές ε, και ε, θέλουμε να τα πονήσουμε το ταχύτερο δυνατό, αλλά σίγουρα έχουμε να κάνουμε εδώ με βάθος ε, των ε, ε, ίσως δύο ετών. Αυτή ήταν λοιπόν η τελευταία μου διαφάνεια και ε, κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το πού βρισκόμαστε. Να σας πω ότι το τέταρτο πακέτο θα υποβληθεί προς ψήφιση από την τεχνική ομάδα ε, την Άνοιξη. Μάρτιο ή Απρίλιο, οπότε δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη διάθεσή μα, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η σωστή διαδικασία αρχέ του επόμενου έτου, το αργότερο από την δική μας γιατι θα πρεπει να ξεκινησει η διαδικασια αρχες του επομενου ετους το αργοτερο απο την τιμή πλευρα και ε, θα γίνει η ψήφιση από κοινού, με, ε, δηλαδή το τέταρτο ε, πακέτο με το WATP, ώστε δηλαδή να μπορεί να τεθεί σε ισχύ από το φθινόπωρο του 2018. Αυτά από την πλευρά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. you very much. Now, το λόγο τώρα για να δούμε ποιος ο κύριος Ντάς Ντάνς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κάποιες ερωτήσεις για την συμμόρφωση, τη συμβατότητα. Το JRC όταν ανάλυσε την, το πέρασμα στην τεχνολογία PEMS μείωσε την ποσότητα που αναμένεται να ποικίλει από το 20% στο 10%. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι πολύ μικρότερος ο παράγοντας συμμόρφωσης. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική βέβαια επιλογή Αυτό όμως θα συνεχίσει να μειώνει ε, να μειώνεται καθώς η τεχνολογία θα βελτιώνεται αυτό το ποσοστό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κάτι πόσο γρήγορα πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στο 1 ε, στο, στον παράγοντα ε, συμμόρφωσης 1. Κάτι άλλο τώρα για τον αριθμό των ε, οικογενειών οχημάτων που θα ελέγχονται από τις εγκρίσεις τύπου. Είναι 30% των οχημάτων της ΗΠΑ, όπως ξέρω, που ελέγχονται από την EPA. Η πρόταση εδώ προλέπει 5%. Εντάξει, το 30% σίγουρα θα μας έδινε ένα πολύ καλύτερο δείγμα. Ποιο είναι το σκεπτικό λοιπόν για το 5%? Ευχαριστώ κύριε Σέκχαουτ. Ευχαριστώ εκτιμούμε ιδιαίτερα την ενημέρωση αυτή για το που βρισκόμαστε. Ε, βεβαίως ε, ε δημιουργούνται κάποια ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, λογικό είναι από τη στιγμή που θα έχουμε τα στοιχεία από τις διάφορες αρχές, από τρίτα μέρη, ότι υπάρχει μια επικύρωση των λεγόμενων δεδομένων. Όμως το θέμα είναι ποιος θα την κάνει αυτή την επικύρωση. Διότι προβλέπω ήδη ότι θα υπάρξουν διάφορες δυνάμεις που δεν θα τους αρέσουν τα στοιχεία από τρίτα μέρη και τελικά θα επιλέξουμε αυτά από τα οποία έχουμε ήδη. Ε, η διαδικασία επικύρωσης δηλαδή είναι και αυτή σημαντική. Όχι να ξεφορτωθούμε δεδομένα τα οποία κάποιοι θέλουν να βλέπουν. Πήγατε κάπως γρήγορα εκεί στο θέμα αυτό της επικύρωσης και το πώς θα λειτουργήσει. Αλλά νομίζω πως είναι κρίσιμο. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι για τα τεστ που θα πρέπει να γίνονται με τα εργαστήρια τα οποία θα είναι επιστοποιημένα. Ε, πόσα όμως εργαστήρια επιστοποιημένα έχουμε στην Ευρώπη. Μήπως είναι πολύ περιοριστικό. Έχει νόημα να είναι επιστοποιημένα βέβαια τα εργαστήρια, αλλά θα ήθελα να ξέρω ε, για τι μεγέθη μιλάμε. Μην επανέλθουμε στους συνήθεις ύποπτους ενδιαφέρον αυτό που είπατε για τις κατευθυντικέ γραμμές για τα defeat devices ε, αλλά υπήρξε ε, ιδιαίτερη κριτική όταν είχαμε την τελική έκθεση ε, της Επιτροπής ε, για τον Dieselgate ε, και εκφραστεί κάποιος ανησυχής για το πώς προσεγγίζουμε αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές. Δηλαδή υπήρχε μια κάποια ευελιξία ε, υπερβολική ευελιξία σε σχέση με τον παράγοντα συμμόρφωσης. Έχει αλλάξει κάτι. Ε, καλό είναι να υπάρχει δεσμευτική νομοθεσία βέβαια, αλλά υπήρχε κάποια βασική κριτική για το πώς λειτουργούν κρατικέ γραμμές. Γενικότερα, μπορείτε να μας πείτε κάτι επ' αυτού. Τι είδους αλλαγές έχουν γίνει. Διότι αν είναι οι ίδιες με αυτές του Ιανουαρίου, τότε πραγματικά θα ανησυχούσα ιδιαίτερα. Και ένα ερώτημα για τα, τα ζητήματα 1, 2, 3 του RDE. Ένα από αυτά είναι τα όρια οδήγησης, driving boundary conditions, συνθήκες συνορίων οδήγησης. Ε, έχουν συμφωνηθεί κάποιες τέτοιες, κάποιες, τέτοια, τέτοιες συνθήκες στο RDE1 και δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και τόσο ακραία αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Σκοπεύετε να αλλάξετε κάτι ε, επ' αυτού, κάτι τελευταίο κάτι που δεν αναφέρθηκε, αλλά υπήρχε στις συστάσεις, στα πλαίσια του Amis, της Επιτροπής για το Dieselgate, και αυτό είναι κάτι το οποίο το έλεγε το EPA και θα κάνουμε τεστ ευνηδιαστικά. Ξέρω βέβαια ότι αυτό είναι κατά του DNA της Ευρώπης, θέλουν να τα ελέγχει όλα, αλλά ε, το καλύτερο είναι να μην ξέρει ε, ο κατασκευαστής ε, πώς θα είναι το τεστ. Διότι κάθε μέρα γίνονται ευνηδιαστικά τεστ από έναν οδηγό στο αυτοκίνητό του. Ε, δεν ακούω όμως, δεν βλέπω πια τίποτα για τα ευνηδιαστικά τεστ. Ε, ενώ είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθούσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτά. Αν θέλετε συνεχίζω, λέει ο κ. Ζέκχαρτ. Ε, λοιπόν, ποιος άλλος θέλει το λόγο. Ωραία. Αυτά. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Λοιπόν, του κυρίου Ντάνς πρώτα τα ερωτήματα. Πότε θα φτάσουμε στον παράγοντα 1 για την συμμόρφωση. Ε, όταν θα, όχι όταν θα ε, νιώθουμε ότι είναι εντάξει τα πράγματα, όχι, όταν θα έχουμε επαρκή στοιχεία. Καταρχήν θα γίνεται ετησίω μια ε, μια αναθεώρηση, ε, μια ανάλυση ετησίω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια σημεία αναφοράς σε σχέση με, τις, με την απόδοση του ΠΕΜΣ θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς λειτουργεί το ΠΕΜ e σε σχέση με ε, τον εξοπλισμό άλλων εργαστηρίων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 15 ε, ο, το ποστό συμμόρφωση. Τώρα μου πείτε αν θα πτάσει το 1 όσοι έχουν τα πράγματα, μάλλον όχι, αλλά ενδεχομένως ε, θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν μπορώ να σα πω όμω τη στιγμή αν θα γίνει αυτό σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Πάντω ο στόχο προφανώ είναι να είμαστε όσο γίνεται πιο ακριβεί σε ό,τι αφορά την απόδοση του BEPS, του, του PEMS, συγγνώμη. Ε, σε ό,τι αφορά τι οικογένειε τώρα, κατά πόσο είναι 30% ή 5% οικογένειε οχημάτων, ναι. Ε, έχουμε διαβρύνει το πεδίο των οικογένειων για την ε, σηματότητα in service, όμως ε, τη συμμόρφωση in service. Τώρα ποιο θα είναι το ποσοστό το οποίο θα, θα ελέγχεται για να είμαστε αξιόπιστοι. Δεν είμαι βέβαιη αν μπορούμε να, να συγκρίνουμε το 5 με το 30% διότι το σύστημα σημαίνει ΗΠΑ είναι κάπως διαφορετικό. Εμείς κάνουμε κάποιες δοκιμές εγκρίσης τύπου ε, και ξαναελέγχουμε το τεστ αργότερα. Ε, δηλαδή έχουμε ένα τεστ τη στιγμή που το αυτοκίνητο ε, τίθεται σε εμπορία. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας αυτή. θα βελτιώσουμε πάντως πιστεύω τη διαδικασία τη έγκρισης τύπου γενικότερα με, αυτό το, με αυτή την πρόταση. Υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα. Το 5% δεν είναι απλά ένα 5% ε, τυχαία. Όχι, γίνεται μια ανάλυση κινδύνου και γίνεται μια επιλογή των οικογενειών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με βάση πληροφορίε που έχουμε εκ των προτέρων. Η αρχή τύπου θα εξετάσει ποιε οικογένειε είναι οι πιο ε, επίφοβες και με βάση αυτό θα γίνει η επιλογή του 5%. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια, ε, ένα σκεπτικό ε, αρκετά ε, ορθολογικό πίσω από αυτό το ποσοστό. Υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα ότι τα τεστ για την έγκριση τύπου ε, κοστίζει, κοστίζουν, ε, είναι επαχθή. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να εξηγήσουμε αυτούς τους αριθμούς, αυτά τα ποσοστά. Τώρα, για τα ερωτήματα του κυρίου Εκχάουτ για την ε, επικύρωση. Πολύ καλό το ερώτημά σας. Και εμείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε ε, ποιος είναι σε καλύτερη θέση για να επικυρώσει τα δεδομένα αυτά τα στοιχεία αυτά για να αποφύγουμε ε, τις καταχρήσεις. Ε, λάβουμε υπόψη μας, παραδείγματος χάρη, τη δυνατότητα να υπάρχει ένα φόρουμ, που, το φόρουμ δηλαδή που υπάρχει ήδη για τη διαδικασία έγκριση τύπου, να το κάνει αυτό το φόρουμ. Ε, υπάρχει και ομάδα πυρογνωμόνων των αρχών έγκριση τύπου, μπορεί να δημιουργηθεί και ένα τρίτο φόρουμ. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστία ε, στην επιλογή αυτή. Δεν μπορώ να σα δώσω μια πλήρη απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά πάντω ε, πραγματικά αναζητούμε το κατάλληλο εργαλείο. Τώρα για, τα, για την πιστοποίηση των εργαστηρίων. Μπορεί να φταίει η διαφάνεια έτσι όπως την έχουμε ε, παρουσιάσει, γίνεται δύο φορές αναφορά στα εγκεκριμένα εργαστήρια. Καταρχήν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν τη δουλειά για, την, για τις αρχές έγκρισης τύπου. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Στα πλαίσια του συστήματος έγκρισης τύπου θα υπάρχει και μια πιστοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών. Ε, αυτό είναι θερμοθετημένο για αυτούς που αποτελούν μέρος του συστήματος έγκρισης τύπου. Τώρα το θέμα είναι τι γίνεται με τα τρίτα εργαστήρια, τα ανεξάρτητα εργαστήρια, πώς θα πιστοποιούνται. Πιστοποιούνται πάντως αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω για πόσα εργαστήρια μιλάμε, πόσα έχουν πιστοποιηθεί, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία να εξελίξει και μόλις έχουμε κάποια νέα στοιχεία θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Ποιος δηλαδή, για το ποιος έχει λάβει αυτή την πιστοποίηση. Για τι κατητήρες γραμμέ τώρα, έπρεπε να ήμουν πιο ακριβή προηγουμένω. Ε, όταν είπα ότι οι κατευθύνσεις γραμμέ ε, θα προχωρήσουν στο τέταρτο IDAC, θα θυμάστε ότι οι κατευθύνσεις γραμμέ αποτελούνται από δύο, δύο σκέλη. Ε, πρώτα απ' όλα τα defeating devices, ε, πώς δηλαδή τα αντιμετωπίζουμε αυτέ τι συσκευέ ε, και πώ τα ερευνούμε και και υπάρχει το θέμα της στρατηγικής ε, εκπομπών. Ε, αυτό το δεύτερο μέρος ε, είναι που θα αποτελέσει μέρος του κειμένου. Γιατί, ε, διότι σκεφτήκαμε ότι πρέπει να εξελίσσονται, εξελίσσονται και τις γραμμές αυτές. Δεν θα ήταν λογικό ε, να τα καταστήσουμε άκαμπτα, να μην μπορούμε να τροποποιήσουμε, να τροποποιήσουμε αυτό το σκέλος κρατητήριων γραμμών. Είναι ένα ζωντανό έγγραφο και μπορώ να σας πω ότι, να σας επιβεβαιώσω ότι βεβαίως να θα λάβουμε υπόψη μας την εμπειρία ε, που θα έχουμε. Καθώ θα αναπτύσσουμε τι κριτέ γραμμέ, λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τι καταστήσουμε πιο ρεαλιστικέ, να αποτυπώνουν, εν περιπτώσει, σαφέστερα, ε, πιστότερα την υπάρχουσα κατάσταση. Τώρα για τα boundary conditions. Δεν θεωρούμε ότι είναι και τόσο ευέλικτα όπω είπατε εσείς ε, αυτά τα όρια, αυτέ τι προποθέσει. Οπότε δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε κάτι επ' αυτού. Κάτι που συνδέεται με το δεύτερο ερώτημα. Τι θα γίνει δηλαδή με τα defeat device και πώς θα αντιμετωπίζουμε. Ό,τι βρίσκεται πέρα από τις συνθήκες ορίων, ε, από τις ωραίες συνθήκες, ε, μας οδηγούν στα defeat devices. Αυτό το περιθώριο 5% θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο. Δεν μπορούμε δηλαδή να ρυθμίσουμε ε, ε, τι συμβαίνει σε εξαιρετικές συνθήκες ε, οδήγησης. Ε, ε, δεν σκοπεύουμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτές τις συνθήκες ε, τις οριακές. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι πώς θα αναζητήσουμε αυτές τις συσκευές, τα defeat devices. Και αυτό είναι το τελευταίο θέμα. Έρχομαι στο τελευταίο θέμα για τους φοινιδιαστικούς ελέγχους. Για την συμβατότητα in service. Αυτό δεν έχει να κάνει με τους αδιαστικού ελέγχους, δεν έχει να κάνει με το να πάμε πέρα από αυτό που προβλέπεται την νομοθεσία. Απλώς αποτυπώνει, ε, αποτυπώνεται το τεστ που έχει προβλέπεται ήδη. Όμω, στο ε, σκέλος που αφορά την εποπτεία της αγοράς, την παρακολούθηση της αγοράς, θα υπάρχει δυνατότητα να πάμε παραπέρα. Πέρα από τα όρια όπως αυτά προβλέπονται ε, για το τεστ ε, συμβατότητας in service. Πιστεύω ότι είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι για να αναζητήσουμε, να εντοπίσουμε ενδεχόμενα defeat devices μέσω της εποπτείας της αγοράς και ξεκινώντας από αυτά που είναι υποχρεωτικά ε, σε επίπεδο θα μπορούμε να πάμε παραπέρα. Όσο έχουν τα εργαλεία σήμερα εμείς ε, θεωρούμε ότι έχουμε περιορίσει όσο γίνεται τις καταχρήσεις. Βεβαίως ε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι βέβαιο και δεν είναι κάτι που θα ισχύει για πάντα. Γι' αυτό λοιπόν θα αναθεωρούμε τακτικά την νομοθεσία. Πιστεύουμε όμως με το σύστημα που θεσπίζουμε, με την έγκριση τύπου, ε, την συμβατότητα in service, την εποπτεία της αγοράς, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα, ε, τα, τα οχήματα θα έχουν την απόδοση που αναμένουμε από αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντάντς. Ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθω στους παράγοντες συμμόρφωσης. Από ό,τι ξέρουμε υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τεχνολογικών δυνατοτήτων. Αναφερθήκατε 0,15 τη διαφοροποίηση όσον αφορά την τεχνολογία PEMS. Αυτό ο βαθμό συμμόρφωσης γιατί είναι ακόμα 2,1. Γιατί πρέπει να περιμένουμε την αναθεώρηση μέχρι ότου να μειωθεί. Δεν θα έπρεπε να έχουμε την περίπτωση κατά την οποία βεβαίω η τεχνολογία πρέπει να αναθεωρηθεί ετησίω, να αναθεωρείται ετησίω. Αυτό είναι λογικό. Αλλά ο παράγων συμμόρφωση αυτό καθ' αν ήδη γνωρίζουμε τεχνολογία, μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν κατανοώ γιατί πρέπει να περιμένουμε. Θέλετε να απαντήσετε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, να υπενθυμίσω κάποια πράγματα. Υπάρχουν δύο παράγοντες συμμόρφωσης. Ένας παράγοντας συμμόρφωσης και ένα περιθώριο. Το 2,1 που αναφέρατε είναι ένας παράγον συμμόρφωσης. Αυτός που συζητήσαμε όλοι τώρα, όσον αφορά τη μείωση της τιμής, είναι περιθώριο. Ο πρώτος, ο τελευταίος μάλλον παράγον, ε, συνδέεται με τον εξοπλισμό, με το PEMS με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδει το PEMS, ενώ το 2,1 Καταρχάς είναι κάτι προσωρινό, θα εξαφανιστεί από μόνο του, από μόνο στο παράγον το 2020-2021, ανάλογα με τα νέα οχήματα τύπου 4 και συνδέεται με στατιστικές αβεβαιότητες μετρήσεως του ΠΕΜ. Δεν σχετίζεται με τον εξοπλισμό, θα θυμόσαστε. Στα πλαίσια του RDI δεύτερο πακέτο, είχαμε τι έντονε αυτέ συζητήσει όπου καθορίσαμε τον παράγοντα συμμόρφωση. Ο πρώτο δεν σχετίζεται με το PEMS. Ε Καθόλου μόνο ο άλλος αριθμός, σύμφωνα το παράδειγμα 2 του RDE, μπορεί να αναθεωρηθεί. Ο πρώτος θα πάψει να υφίσταται τον Ιανουάριο 2020 για τύπους ε, και το 2021 για όλα τα χήματα. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Καλώς, μέχρι τότε. Σας ευχαριστούμε για την ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος. Πάμε στο επόμενο σημείο τη διάταξης. Ερωτήσεις για τον κανονισμό, το σχετικό με ενημέρωση των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα και πληροφορίες που χορηγούνται στους καταναλωτές. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και την ενημέρωση τρόφιμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Αλεξάνδρα Νικολοκοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας, Σάντε, είναι εδώ. Μπορείτε να κάνετε ένα νεύμα, αν είστε εδώ, παρακαλώ. Α, δεν είναι, δεν ήρθε ακόμα. Μπορεί να μας πει κάποιος κάτι από πλευράς Κομισιόν. Θα περιμένουμε να καταφτάσει η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπετε, προχωρήσαμε πιο γρήγορα, είμαστε ένα δεκάλεπτο πιο νωρίς από ό,τι προβλεπόταν. Περιμένουμε ένα δεκάλεπτο, λοιπόν. Την κυρία Νικολακοπούλου. Να έρθει η κυρία Νικολακοπούλου. Και μετά θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Everyone, thank you. <laughs> Um, so, dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε λοιπόν στο σημείο της σημερινής διάταξης. Ερωτήσεων αφορά την παροχή πληροφοριών τα τρόφιμα στους καταναλωτές, κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Θα ακολουθήσουμε τη σειρά τους σύμφωνα τις διατάξεις του κανονισμού. Ομαδο, θα ομαδοποιηθούν. Κατά θέματα. Για κάθε θέμα θα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στα μέλη για ερωτήσει: σχόλια, παρατηρήσεις, θεμητές πρακτικές πληροφόρησης και ενημέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει και έχει το λόγο. Ορίστε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας που με απευθύνθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Έτσι μπορούμε να κάνουμε επισκόπηση της καταστάσεως όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για την ενημέρωση για τα τρόφιμα. Τα ερωτήματα καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων. Καταρχάς, η κυρία Γκέρλινγκ, ερώτηση θεμητές πρακτικές ενημέρωσης. Ρωτά, κάποιες ετικέτες που υπάρχουν στην αγορά τώρα, όπως για ε, το έλαιο, το φινικέλαιο, που λέει ότι είναι ελεύθερο από κάποιες ουσίες, free from θα πρέπει να είναι σαφής, σαφές ότι η ενημέρωση, η απουσία στατικών από κάποια τρόφιμα μπορεί να παρέχεται εθελοντικά από επιχειρηματίες και πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις πληροφορίες που παρέχονται εθελοντικά. Άρθρο 36 του κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες που χορηγούνται εθελοντικώς δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφισημία, να μην επικρατεί σύγχυση, να δημιουργείται σύγχυση. Και όπου ενδείκνεται πρέπει να βασίζεται επί των συγκεκριμένων σχετικών επιστημονικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό, 7.1.C 7.1c, οι πληροφορίε στα τρόφιμα θα ήταν παραπλανητικές εάν ισχυρίζονται ότι το τρόφιμα κατέχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όταν όλα παρόμοια τρόφιμα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά τονίζοντας ιδιαίτερα την παρουσία ή την απουσία κάποιων συστατικών. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για το φινικέλαιο που είναι ελεύθερο από προϊόντα που εν πάση περιπτώσει δεν χρησιμοποιούν. Α, για ένα προϊόν που δεν έχει φινικέλαιο ε, δεν συμμορφώνεται, δεν ταιριάζει με αυτή την απέτηση. Βασική αρχή. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή της νομοθεσίας και για την εξακρίβωση κατά πόσο η ετικετοθεσία συνάδει με το εφαρμοστέο δίκαιο. Πιστεύουμε ότι οι ισχύοντες κανόνες ήδη παρέχουν τα αναγκαία εχέγγυα για να προστατεύονται οι καταναλωτές από παραπλανητικές πληροφορίες και συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φρονεί ότι απαιτείται να προστεθούν άλλα μέτρα στον τομέα αυτό. Σχόλιο υπάρχει. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Συνεχίζοντας. Το άρθρο 36 δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το συγκεκριμένο και ξεκάθαρο. Δεν γνωρίζω να έχουν δρομολογηθεί δράσεις και προσφυγές βάσει το άρθρο 36. Ξέρω όμως ότι πολλά προϊόντα διατίθεται στην αγορά που παραβαίνουν το λόγο άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποιεί τις οδηγίες που δίνει στα κράτη-μέλη. διότι εν ώψη του πολλαπλασιασμού των νέων προϊόντων που παραπλανούν τους καταναλωτές και θα έχουν παραπλανητικές ετικέτες σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνει κάτι να αντιταχθεί σε αυτή την τάση. Μπορεί να το εξετάσει αυτό. Να στείλει κάτι, να ειδοποιεί τα κράτη-μέλη γι' αυτό ότι ενδεχομένω θα μπορούσε αυτό το πλαίσιο να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 36. Μπορείτε να απαντήσετε. κάποιος άλλος. Όπως σας είπα, υπάρχουν δύο διατάξεις που είναι σχετικές με το θέμα. Η μία το άρθρο 36 που πράγματι προβλέπει γενικά κριτήρια. Δεν είναι σωστός ο κατάλογος βέβαια, σωστά το λέτε. Είναι θέμα αξιολογήσεως από τις αρμόδιες αρχές. Τι είναι παραπλανητικό ή όχι, τι είναι αμφίσιμο ή όχι, όμως αυτό θα πρέπει να ερμηνευθεί σε συνάρτηση με το άλλο άρθρο που αναφέρεται στην ερώτηση. Το 7.1 γάμα, όπου εκεί σαφώς αναφέρεται ότι είναι παραπλανητικό να αναφέρει κανείς την απουσία συστατικού ή να τονίζει την παρουσία ενός συστατικού όταν αυτό ισχύει για όλα τα άλλα παρόμοια προϊόντα. Αν τονίζοντας την απουσία ενός συστατικού, δημιουργείται εντύπωση για τον καταναλωτή ότι αυτό το τρόφιμο έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτό σαφώς είναι κάτι παραπλανητικό. Εδώ λοιπόν έχουμε σαφή κριτήρια, τα οποία μαζί με το 36 μπορούν να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες αρχές. Γενικότερα τώρα εάν ξεπεράσουμε αυτά τα παραδείγματα, εάν κάποιο προϊόν δεν έχει κάποιο στατικό ή περιέχει κάποιο στατικό, πράγματι το άθρο 36 είναι γενικό λόγο. Δεν μας ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να παράσχουμε συγκεκριμένο προσανατολισμό επ' αυτού. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι μέχρι τώρα η πρακτική ποια είναι. Όταν έχουν συγκεκριμένα προβλήματα που ένα κράτος μέλος χρειάζεται κάποια συμβουλή και προσανατολισμό, το θέτει στο φόρουμ συζητήσεως είτε στη μόνιμη επιτροπή, στη διευθύνουσα επιτροπή ή στην ομάδα εργασίας για την ετικοτοθεσία και καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πρακτικά συγκεκριμένες πρακτικές που μπορεί να θεωρηθούν ως παραπλανητικές. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτή τη φάση δεν προτιθέμεθα να εκδώσουμε γενικούς προσανατολισμούς σχετικά με την εφαρμογή του άθρου 36. Ευχαριστώ. μπορούμε να προχωρήσουμε. Επόμενο θέμα. Πόσο ευανάγνωστα είναι τα, πώς ευανάγνωστα είναι το μέγεθος των γραμματοσυρών με άλλα λόγια. Ευχαριστώ. Εδώ η ερώτηση αναφέρεται σε ένα θέμα που συζητήθηκε εκτενώς Πώ ευανάγνωστες είναι ετικέτε με του συνομοθέτε συζητήθηκε για να υιοθετηθεί ο κανονισμός. Μετά από πολλές συζητήσει. συμφωνήσαμε ότι οι πληροφορίες στα τρόπιμα πρέπει να είναι ευανάγνωστες, αδιαφυσβήτητο αυτό, και ποια ήταν η απόφαση. Να καθορίσουμε το τι είναι ευανάγνωστο. Κάτι ευανάγνωστο εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των γραμμάτων, το είδος γραμματοσυράς και το μέγεθος αυτής και γενική η παρουσίαση των πληροφοριών, των υποχρεωτικών, πώς γίνεται, για να είναι ανάγνωστη ετικέτα. Ελάχιστο μέγεθος, ε, καθορίστηκε για τη με κάποια ευελιξία για μικρές συσκευασίε. Όπως δείχνει και το παράδειγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα εύκολο να εξασφαλίζεται το ευανάγνωστο της ετικέτας, κυρίως στις μικρές συσκευασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείε τροφίμων προσπαθούν να συμπεριλάβουν αρκετές γλώσσες στην ετικέτα. Η ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μπορούμε να εξετάσουμε τον δεχόμενο να χρησιμοποιούμε αντί της ετικέτας άλλους τρόπους παροχής των λόγω πληροφοριών σε συσκευασμένα τρόφιμα. Τώρα, σύμφωνα με τον κανονισμό και αυτά που ισχύουν τώρα, Πρέπει να πούμε ότι οι υποχρεωτικέ αυτέ πληροφορίε πρέπει να παρασχόνται, πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα στη συσκευασία ή σε ετικέτα που είναι επικολλημένη. Αυτό είναι ο κανόνα. Τι σημαίνει αυτό. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική ετικέτα ούτω υπήν δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν να παρέχονται επιπλέον πέραν της ετικέτας της βασικής. Τώρα αν αυτός ο κανόνας θα πρέπει να αλλάξει ούτως ώστε να επιτρέπεται μία άλλη μέθοδος παροχής των πληροφοριών. Αυτό είναι ένα θέμα προς εξέταση. Να σας υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός για την ενημέρωση των φατατρόφιμα παρέχει τη δυνατότητα, υπάρχει η πρόβλεψη στον κανονισμό, η δυνατότητα χρησιμοποίησης διαφορετικών τρόπων πληροφόρησης. Αυτό πρέπει να γίνει σε δύο στάδια. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει καταρχάς με καταξισοδότηση πράξη ποια θα είναι τα κριτήρια για κάτι τέτοιο και αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί από εφαρμοστική πράξη. Αυτό είναι εφικτό και αυτό θα απαιτούσε μία αλλαγή των ισιών των κανόνων. Με τους ισχύοντες κανόνες αυτό δεν επιτρέπεται. Ευχαριστώ. Ποιος έχει κάτι να πει. Ο κύριο Τόλιτς. Όχι. Ναι. Ο κύριο Τόλιτς είχε θέσει το ερώτημα και γι' αυτό τον ρώτησα. Α, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω κρατικά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν τεθεί ερωτήσεις. Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω οι συμπληρωματικές πληροφορίες, κυρίως όσον αφορά τον ευανάγνωστο χαρακτήρα της ετικέτας, είναι θέματα που αναφέρθηκαν. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Πέρα από τις υποχρεωτικές πληροφορίες και την υποχρεωτική ετικετοθεσία, θα ήταν καλό να χορηγούνται συμπληρωματικέ πληροφορίε στου καταναλωτέ σχετικά με την προέλευση ενό προϊόντο, σχετικά με τα στατικά του προϊόντο κλπ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ ένα ερώτημα, το οποίο δεν αναφέρθηκε εδώ, αλλά το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα που συζητούμε τώρα. Ο κανονισμός προβλέπει ότι η Επιτροπή παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά περαιτέρω κριτήρια, σε ό,τι αφορά ε, το ευανάγνωστο αυτών των υποχρεωτικών πληροφοριών. Χωρί όμω να υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο. Δεν έχει τεθεί δηλαδή εδώ προθεσμία. Οπότε αυτό που θέλω να ακούσω από την Επιτροπή είναι είναι διατεθειμένη να εκπονήσει περαιτέρω κριτήρια σε ό,τι αφορά το επανάγνωστο αυτών των στοιχείων επάνω στην σήμερα, Δηλαδή αναφέρομαι εδώ στη γραμματοσυρά, την απόσταση των χαρακτήρων μεταξύ του, το μέγεθο των χαρακτήρων και ούτω καθεξής. Μία σειρά δηλαδή από διαφορετικά κριτήρια τα οποία θα μπορούσαν και μπορούν να συμβάλλουν ε, στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας ε, των πληροφοριών. Ε, και εδώ το θυμίζω και στου συναδέλφου που ενδεχομένω κάποιοι να το θυμούνται από την προηγούμενη ε, τη θητεία, ε, το ευανάγνωστο, αν θέλετε, αυτή η αναγνωσιμότητα δεν ε, ορίζεται ω τέτοια. Οπότε θα πρέπει να ε, οριστούν ορισμένα κριτήρια. Αλλά όταν είχαμε κάνει τον τριμερή διάλογο, είχαμε καταλήξει μόνο στο μέγεθο τη γραμματοσυρά και σε τίποτα άλλο. Και γι' αυτό η Επιτροπή τότε είχε πει ότι ήταν διατεθειμένη να εξετάσει περαιτέρω κριτήρια σε ό,τι αφορά ακριβώ την αναγνωσιμότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει το λόγο. Η κυρία Σόμερ έθεσε το γενικότερο ερώτημα. Όσον αφορά τι υποχρεώσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι λογικό να καλυφθεί από αυτό το συγκεκριμένο σημείο, το ειδικό. Να πω λοιπόν ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το βλέπει το θέμα αυτό ως θέμα προτεραιότητας για να υιοθετηθούν συμπληρωματικοί ε, κανόνες για την αναγνωσιμότητα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναγνωρίστηκε ότι η αναγνωσιμότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος των χαρακτήρων της γραμματοσυράς και γι' αυτό λάβαμε υπόψη την τροπολογία του Ευρωκοινοβουλίου. Συμπεριλήφθηκε ο ορισμός του ευανάγνωστου της ετικέτας, πέρα της αρχικής προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλάβαμε το μέγεθος των χαρακτήρων συν ορισμό της αγνωσιμότητας, του ευανάγνωστου της ετικέτας που εμπεριέχει και άλλα κριτήρια. Τι σημαίνει στην πράξη. Αν μια ετικέτα τροφή μου, αν συμμορφώνεται με το ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμμορφούνται με την απέτηση να είναι βανάγνωστη ετικέτα διότι οι ελεγκτές των τροφίμων θα πρέπει να λάβουν υπόψη και άλλα κριτήρια. Παραδείγματο χάρη, έχουμε μια ετικέτα που σέβεται το ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων, αλλά με την αντίθεση, με το κοντράστ μεταξύ χρωμάτων και ετικέτας δεν είναι ευανάγνωστη ετικέτα, τότε βάσει του ορισμού του ευανάγνωστου του, της ετικέτας, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν είναι ευανάγνωστη ετικέτα Πράγματι, δεν έχουμε προχωρήσει τόσο μακριά να καθορίσουμε ποιος θα, ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ των γραμμών ή η απόσταση μεταξύ των ε, χαρακτήρων. Ε, πιστεύουμε παρόλα αυτά ότι υπάρχουν τρόποι ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι ετικέτες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να επιβάλλονται κυρώσεις που στρέφονται κατά των πρακτικών που δεν συμμορφώνονται με την απέτηση για ευανάγνωστες ετικέτες. Και πιστεύουμε ότι θα ήταν λογικό να γίνει μια αξιολόγηση του πώς οι ισχύοντες κανόνες εξασφαλίζουν ευανάγνωστες ετικέτες και μετά να ακολουθήσουμε με θέσπιση συμπληρωματικών κανόνων. Θέλουμε να δώσουμε κάποιο χρόνο στον κανονισμό αυτό, να μας δώσει κάποια αποτελέσματα και μετά να κάνουμε αξιολόγηση και βλέπουμε Υπέρχουμε νομική υποχρέωση και πρέπει να το επαναξετάσουμε, αλλά δεν είναι θέμα που έχει προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Τρίτο θέμα. Κατάλογο συστατικών υλικού και εφαρμογή ε, της, ε, του κανονισμού για ε, τις πολύ μικρές ετικέτες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Οι τρεις ερωτήσεις αναφέρονται όλες στους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί σε τέσσερα κράτη-μέλη. Γαλλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία το 2017 για την ετικετοθεσία των τροφίμων. Πράγματι, η έκθεση που σχετίζεται με τους διενεργηθέντες ελέγχους στη Γαλλία αναφέρεται και σε πορίσματα που αφορά ε, νάνο ετικετοθεσία. Άλλες τρεις χώρες, στις σχετικές εκθέσεις της χώρες, δεν εμπεριέχονται στοιχεία όσον αφορά τη συμμόρφωση με, το, ε, με την ετικετοθεσία και την αναφορά νάνο συστατικών. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων ήταν τέτοιος που είχε στόχο την κάλυψη των στόχων, <laughs> συγγνώμη, την κάλυψη των ε, προδιαγραφών, αν υπάρχει συμμόρφωση. Ήταν ευρύ το πεδίο των ελέγχων. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τις ελεγκτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εστιαστήκαμε επί κάποιων πτυχών του κανονισμού. Θυμάμαι ε, τα αλογόνα, ε, ημερομηνία λήξης, διατροφικές ιδιότητες και χώρα παραγωγής προέλευσης. Ε, εκεί είχαμε ζητήσει να επικοινωθούν οι έλεγχοι. Το ότι υπάρχουν πληροφορίες για τα ανών συστατικά στη γαλλική έκθεση, αυτό οφείλεται σε ίδια πρωτοβουλία. Η Γαλλία έθεσε το ζήτημα από μόνη της στα πλαίσια ενός προγράμματος γαλλικού. Τώρα, θέλουμε να κάνουμε και νέους ελέγχους το 2018 σε τέσσερα κράτη-μέλη και πάλι. Και υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το θεωρεί ότι ενδείκνυται, να θέσει στόχους Συγκεκριμένου. που αφορούν συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού. Θα μπορούσαμε να δώσουμε έμφαση και στην ετικητοθεσία όσον αφορά τα νάνο συστατικά. Ωραία. Ερωτήσεις. Όχι. Επόμενο θέμα. Χώρα προέλευσης ή τόπος προέλευσης, χώρος προέλευσης. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Τέσσερις τα σχόλιά σας όσον αφορά τις ερωτήσεις και μετά θα δούμε εάν θα υπάρξουν και άλλα ερωτηματικά. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις είχαμε. Της κυρίας Ζόμερ και του κυρίου Παουλούτσι όσον αφορά την εφαρμοστική πράξη που αφορά ε, την δικαιοθεσία ε, προέλευσης, αφορά της προέλευσης και σχετίζει την έγκριση, την υιοθέτηση του κανονισμού με τα εθνικά μέτρα όσον αφορά την ε, αναφορά της χώρας προέλευσης. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνουμε τις εσωτερικές διεργασίες. Συζητήσαμε εκτενώς το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μαζί με τα κάτι μέλη το κουβεντιάσαμε. και θεωρούμε ότι έχουμε καταλήξει κάποια συμφωνία. Αυτό τι σημαίνει. Ότι συντομότατα θα έχουμε έτοιμο ένα σχέδιο κειμένου που θα δημοσιευθεί στην πύλη για την καλύτερη νομοθεσία για να υπάρξει κάποια αντίδραση. Ακολουθούμε τους κανόνες για την καλύτερη θέσπιση νομοθεσίας. Κοινοποιούμε όλα αυτά τα κείμενα στους εμπορικούς εταίρους, στον ΠΟΕ, και μετά θα υποβληθεί το θέμα στα κράτη-μέλη, στη Ρυθμιστική Επιτροπή, στην ε, Μόνιμη Επιτροπή, ελπίζοντας ότι θα πετύχουμε μια ειδική πλειοψηφία. Σύμφωνα με το σχέδιό μας λοιπόν, πιστεύουμε λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα βήματα της διαδικασίας, πιστεύουμε λέγω ότι ο φορμαστικός κανονισμός θα το πρώτο εξάμεινο του 2018. Βέβαια, αν φτάσουμε ε, στην ειδική πλειοψηφία, να συλλέξουμε την ειδική πλειοψηφία, να αναφερθώ σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την, ονομασία, την ε, αναφορά της προέλευσης του προϊόντος, νομίζω τα κάλυψα. Ο κ. Καπούτο και η κυρία Γιατενμάκη έκανα κάποια ερώτηση. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν το θέμα που υθετήθηκε το 2016 και ζητήθηκε μία επέκταση ε, της υποχρετικής αναφοράς ε, προέλευσης να καλύπτει και άλλα προϊόντα. Και ερώτηση είναι ποια συνέχεια δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω κάτι. Έχουμε κάνει κάποια εργασία πάνω σε αυτό το θέμα όσον αφορά την ετικετασία προέλευσης Υιοθετήσαμε διάφορες εκθέσεις που ζητήθηκαν από τον κανονισμό να δούμε τη δυνατότητα να θεσπιστεί υποχρεωτική αναφορά χώρας προέλευσης ή τόπου προέλευσης για κάποιες κατηγορίες τροφίμων όπως συστατικά γάλακτος, ε, μη καταργασμένα προϊόντα, προϊόντα με ένα συστατικό και προϊόντα που έχουν πάνω 50% ενός συστατικού στο τρόφιμο, υιοθετήθηκαν όλα το μόνο που εκκρεμεί οφάσεις νομικές νομικέ υποχρεώσει είναι αυτή η εφαρμοστική πράξη όσον αφορά την κοιτοθεσία προέλευσης. Και τρεις εκθέσεις που υιοθετήσαμε καταδεικνύουν, όπως είπαμε πανηλημμένα, ότι η υποχρεωτική κοιτοθεσία προέλευσης για διάφορα προϊόντα σχετίζεται μάλλον έχει αντίκτυπο σημαντικό που μπορεί να αυξήσει το διοικητικό άχθος και να επηρεάσει το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το αναφέραμε και στην απάντησή μας στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Λοιπόν, τι είχαμε πει και το επαναλαμβάνουμε, ότι προτιμάμε εθελοντική ετικετοθεσία προέλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ο καταναλωτής μπορεί να διαλέξει προϊόντα με συγκεκριμένη προέλευση, αν θέλει να το κάνει αυτό, ενώ δεν επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα των διαφόρων εταιριών τροφίμων. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα κρατη Γαλλία, Ιταλία, η Λιθουανία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία ήδη έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν πειραματικά εθνικά προγράμματα στον τομέα αυτό όπως το έχουν αποκαλέσει και έχουν θεσπίσει υποχρεωτική αναφορά για ε, γάλα ε, προϊόντα γάλακτος και προϊόντα κρέατος και οι χώρες πριν το τέλος της δοκιμαστικής περίοδου της, ε, του εθνικού πειραματισμού θα υποβάλλουν έκθεση όσον αφορά τη λειτουργία που έχει το σύστημα και τι αντίκτυπο έχει στην εσωτερική αγορά. Βάσει των νέων στοιχείων τα οποία θα ολοκληρώσουν τα απορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τα απορίσματα που θα συλλέξουμε από τους ελέγχους που διενεργούνται σε κάποια κάτι μέλη. Με όλα αυτά θα αξιολογήσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω αν χρειάζεται να διαρευνήσουμε για δίποτε νέα πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως επ' αυτού. Και μετά έχουμε μια τελευταία ερώτηση για την εκθεσία προέλευσης, πιο συγκεκριμένη. Ο κ. Στόλικα, στο ερώτημα αναφορά χώρας προέλευσης για ομοιογενείς ουσίες, προϊόντα που παράγονται σαν αποτέλεσμα ανάμιξης δύο ή περισσότερων ταυτοσύμων προϊόντων διαφορετικής προέλευσης. Να διευκρινίσουμε κάτι. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι πληροφορίες προέλευσης πρέπει να χορηγούνται πάντα αν η μία αναφορά παραπλανά τον ε, καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική προέλευση του τρόφιμου. Αυτό ισχύει για όλα τα τρόφιμα, είτε είναι ομοιογενή είτε ετερογενή. Ο κανονισμός για την ενημέρωση αφορά τα τρόφιμα για πρώτη φορά προβλέπει ότι η χώρα προέλευσης ενός τροφίμου καθορίζεται σύμφωνα με τους τελωνιακούς κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δηλαδή, για τρόφιμα, η παραγωγή των οποίων συνεπάγεται πάνω από μια χώρα, εμπλέκεται μια, πάνω από μια χώρα, η χώρα προέλευση αντιστοιχεί αντί αυτή η περιπτώση στον τόπο τελευταία ουσιαστική μεταποίηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει κάποια κριτήρια και υπάρχει καταξισοδότηση πράξη σύμφωνα με τον Τελεινικό Κώδικα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και σχετικό κανονισμό αξιολογώντας τι θεωρείται σαν τελευταία ουσιαστική μεταποίηση για τους σκοπούς της αναφοράς, της ανάθεσης μιας προέλευσης σε ένα τρόφιμο, σε ένα προϊόν. Τώρα, κατά πόσο οι πληροφορίε στον φατή χώρα προέλευσης παρέχονται σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια και κατά πόσο αυτό είναι κάτι παραπλανητικό, αυτό αξιολογείται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαφορετικές φάσεις παραγωγής του τρόφιμου. Κάποια τρόφιμα, και τώρα αναφέρομαι στα παραδείγματα που περιέχει η ερώτηση, όπως ε, το μέλι και το ελαιόλαδο, κάποια προϊόντα υπόκεινται σε συγκεκριμένη νομοθεσία ε, όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα για την αναφορά της χώρας προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα. Όσον αφορά το ελαιόλαδο, Εάν υπάρχουν διάφορες χώρες οι οποίες εμπλέκονται στο προϊόν, η ένδειξη θα μπορεί να είναι πιο ευέλικτη. Να λέει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένδειξη να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, EU. Η δεμή, όλες οι χώρες θα πρέπει να αναφέρονται. Παρομοία είναι η κατάσταση και για το μέλι. Και το μέλι καλύπτεται ευελιξία. Αν δεν είναι μια χώρα παραγωγής που εμπλέκεται, η μόνη ευελιξία που παρέχεται στον κανονισμό είναι ή να γράφει EU ε, το μέλι ή ό, όχι EU. Αλλά να μίξεις τώρα ελληνικό μέλη με ιταλικό μέλι και σύμφωνα με τα ποσοστά αν το ελληνικό μέλι είναι 70% και η εταιρεία αποφασίσει να αγνοήσει το ιταλικό μέλι και πει ότι είναι ελληνικό μέλι, ε, εν αυτή η περιπτώση αυτό δεν συνάδει με τον κανονισμό. Λοιπόν, είτε όλες οι χώρες θα πρέπει να αναφέρονται στο προϊόν, είτε προβλέπεται η ευελιξία στον κανονισμό, θα λέει EU ή non-EU στην ετικέτα. Αλλά αναφέρεται μία χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αναμειγνύονται και άλλε, τότε αυτό είναι παραπλανητικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν προτίθεται να υιοθετήσει συμπληρωματικά μέτρα άλλα, διότι πιστεύουμε ότι οι ισχύοντε κανόνε ήδη καλύπτουν τι αναφερόμενε ανησυχίε που συμπεριλαμβάνονται στο ερώτημα του, ειρητή μου βουλευτού. Okay, then thank you for your answers. We move to additional forms of expression. Ναι. Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές ε, ε, πληροφορίες και τις ε, συμπληρωματικές μορφές έκφρασης αυτών των πληροφοριών, υπάρχουν κάποια συμπληρωματικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Μπορείτε να ξεκινήσετε αν θέλετε. Yes, thank you very much. Ε, ναι, σας ευχαριστώ. Η κυρία Σόμερ, ο κύριος Παολούτσι και ο κύριος Στάις έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με αυτό το σημείο. Α, όλα αυτά λοιπόν τα ερωτήματα αναφέρονται στο πού βρισκόμαστε σε σχέση με την έκθεση την οποία θα πρέπει να έχει υιοθετήσει η Επιτροπή στα τέλη του 2017 σε ό,τι αφορά τις συμπληρωματικές μορφές έκφρασης και ε, παρουσίασης της δήλωσης διατροφικής αξίας ή διατροφικών πληροφοριών. Θα δώσω λοιπόν μία απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα μαζί, διευκρινίζοντας καταρχήν το κατά πόσο η Επιτροπή θα εξετάσει το Nutri-Score, αυτό δηλαδή το πρόσφατο σύστημα που θέσπισε η Γαλλία ε, και το καθεξής. Θα ήθελα λοιπόν να σας εξηγήσω ότι ε, τη σήμερα ημέρα τα, τα μόνα συστήματα που υπάρχουν και λειτουργούν στην αγορά και τα οποία πληρούν ή όχι πληρούν ή θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως συμπληρωματικοί τρόποι ε, ε παρουσίασης αυτών των διατροφικών πληροφοριών είναι το Traffic Light ε, του το Ηνωμένου Βασιλείου και το σύστημα GDA το οποίο ήδη αποτελεί τμήμα της νομοθεσίας. Αυτά λοιπόν αποτελούν συμπληρωματικούς τρόπους έκφρασης και παρουσίασης των διατροφικών πληροφοριών. Υπάρχουν τώρα, αυτή την περίοδο δηλαδή, συστήματα τα οποία σχεδιάζονται, όπως το γαλλικό Nutri-Score, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, αξιολογήσει ως σύστημα του άρθρου 35. Θεωρεί δηλαδή πως αποτελεί εθελοντικές συμπληρωματικές πληροφορίες. Και από εκεί και μετά υπάρχει ένα σύστημα το οποίο συζητείται αυτή την περίοδο από έξι πολυεθνικές εταιρείε από το χώρο των τροφίμων και το οποίο όμως δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί. Υπάρχουν επίσης στην αγορά άλλα συστήματα τα οποία στοχεύουν ακριβώς στην παροχή απλούστερων, σαφέστερων πληροφοριών στο καταναλωτή σε ό,τι αφορά ε, τα διατροφικά συστατικά. Το προφίλ, αν θέλετε, διατροφικό, το διατροφικό χαρακτήρα, αν θέλετε, του προϊόντος όπως το σύστημα Keyhole, το σκανδιναβικό αυτό σύστημα. Αλλά και πάλι τέτοιου είδους συστήματα δεν θεωρούμε πως είναι συστήματα που καλύπτονται από το άρθρο 35. Αυτά λοιπόν τα συστήματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καονισμού κανονισμού σε ό,τι αφορά τα health claims, τη δηλώση σε σχέση με την υγεία. Θεωρούμε λοιπόν από την πλευρά της Επιτροπής ότι προκειμένου να επονήσουμε μία πλήρη έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει ε, και μία αξιολόγηση του αντικτύπου αυτών των συστημάτων θα πρέπει το ε, πεδίο που θα καλύψει αυτή η έκθεση να διευρυνθεί έτσι ώστε να μην καλύπτει μόνο αυτά τα δύο συστήματα που θεωρούμε πως επίπτονται στο 35. Προκειμένου με άλλα λόγια να καλύπτει δηλαδή και άλλα συστήματα όπως αυτά που ανέφερα μόλις τώρα το γαλλικό Nutri-Score, το Keyhole System των οπτικών. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το σύστημα των traffic light του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία κατά παράβαση μετά από μία σειρά από αναφορές, από καταγγελίες δηλαδή που έγιναν και αυτό σημαίνει ότι όσο ακόμα τρέχει αυτή η διαδικασία κατά παράβαση θα είναι δύσκολο η Επιτροπή να αποκαλύψει μια σειρά από πληροφορίες και στοιχεία σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο αυτού του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν το, ε, το λόγο αποφασίσαμε να αναβάλουμε την υιοθέτηση αυτής της έκθεσης έω τα τέλη του 2018 ελπίζοντας ότι στο ενδιάμεσο διάστημα θα έχουμε συλλέξει περισσότερα στοιχεία, περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των υφιστάμενων αυτών συστημάτων. Στον διάμεσο διάστημα, η Επιτροπή ζήτησε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το JRC, να προβεί σε μια εκτενή εξέταση της σχετικής βιβλιογραφίας σε ό,τι αφορά ε, τις ε, ε διαφορετικές αυτές ε, μορφές των ε, συστημάτων για τις διατροφικές πληροφορίες. Μία τέτοια λοιπόν εξέταση βιβλιογραφία από το JRC θα μα επιτρέψει να λάβουμε υπόψη μα καλύτερα τον αντίκτυπο αυτών των συστημάτων στην δική μα έκθεση. Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχει και μια αξιολόγηση στο πλαίσιο του REFIT του κανονισμού κατά υγείας και από αυτήν λοιπόν την διαδικασία REFIT θα λάβουμε και χρήσιμε πληροφορίε και από τον ανάδοχο τη σχετική μελέτη καθώς εκείνος θα εξετάσει και τα συστήματα αυτά, δηλαδή των εναλλακτικών συστημάτων έκφρασης των σχετικών πληροφοριών. Παρότι λοιπόν έχουμε ξεκινήσει την όλη διαδικασία, είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να σας ε, παράσουμε πληροφορίες στο τι είδους πορίσματα θα περιλαμβάνει η εν λόγω έκθεση. Μόνο όταν δηλαδή θα έχουμε ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες που ανέφερα μόλις τώρα, θα είμαστε σε θέση να σας πούμε κατά πόσο υπάρχει πράγματι ανάγκη θέσπισης εναρμονισμένων κριτηρίων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως πέραν αυτών των ερωτημάτων τέθηκε και ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά το άρθρο 36 παράγραφος 3 ή μάλλον 36 παράγραφος 4 διορθώνει η ομιλήτρια το οποίο προβλέπει η Επιτροπή θα πρέπει να καθετεί κατεξοδότηση πράξη σε ό,τι αφορά άλλες εθνολωτικέ πληροφορίες. 36-3 λέει τώρα μιλήτρια. Ε, το 36 λοιπόν 3 προβλέπει τη δυνατότητα ευθέτηση κατεξοδότηση πράξεων για την Επιτροπή σε ό,τι αφορά πρωτοτυπικέ πληροφορίε ή σε ό,τι αφορά τρόφιμα για φυτοφάγου και για vegans αλλά και σε ό,τι αφορά δεδομένα για συγκεκριμένε ομάδε του πληθυσμού. Το ερώτημα λοιπόν που τέθηκε ήταν, σκοπεύει πράγματι η Επιτροπή να υιοθετήσει περαιτέρω κατεξοδότηση πράξη έτσι ώστε να εναρμονίσει τα κριτήρια για άλλου είδου ε, πληροφορίε. πληροφορίες. Η απάντησή μας λοιπόν είναι ότι δεν σκοπεύουμε αυτή τη στιγμή να το κάνουμε, αλλά εάν ανακύψει μια σχετική ανάγκη θα το πράξουμε. Όμως προς το παρόν δεν έχουμε ε, αναγνωρίσει κάποια ανάγκη για την υιοθέτηση τέτοιου είδους συμπληρωματικών κανόνων ε, ε, και το τομέων σε ό,τι αφορά αυτές τις συμπληρωματικές εθνωτικές πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παραγραφός 3. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Σχόλια σε σχέση με αυτό το σημείο. Η κυρία Ζόμερ έχει το λόγο. Ναι, ε, είμαι έκπληκτη από το γεγονός ότι η Επιτροπή θεωρεί πως ε, με όλα αυτά τα νέα συστήματα που προκύπτουν σε εθνικό επίπεδο δεν χρήζουν κάποιες δράσεις. Καθώς αυτός ο τομέας αποτελείται κατά 90% από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα μπορούν να είναι βέβαιες για το τι ισχύει στα άλλα κράτη-μέλη, ώστε να είναι σε θέση να εξάγουν σε αυτά τα άλλα κράτη-μέλη Ειδικότερα όταν η Επιτροπή μας λέει ότι ένα εθνικό σύστημα όπως το ε, Nutri-Score ε, ούτε καν εμπίπτει στο άρθρο 35 και κατά συνέπεια ε, δεν υπάρχει ζήτημα. Μα δεν πρόκειται ουσιαστικά για ένα υποχρεωτικό σύστημα που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο σε αυτή την περίπτωση. Και δεν μπορούν να παρεύουν και άλλες γενικές διευθύνσεις. Δηλαδή Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τη αγορά. Ε, και ποιο ήταν ο στόχο του κανονισμού. Ακριβώ να ενοποιήσουμε, να εναρμονίσουμε μεταξύ του όλα αυτά τα συστήματα ε, των πληροφοριών, ακριβώ για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε ό,τι αφορά την εμπορική δραστηριότητα. Και θα ήθελα ε, να γνωρίζω κατά πόσο η Επιτροπή έχει εξετάσει και το επιστημονικό υπόβαθρο αυτών των εθνικών συστημάτων που έχουν αρχίσει να ανακύπτουν, γιατί κάτι τέτοιο προβλέπεται άλλωστε στον κανονισμό ή απλά η Επιτροπή λέει «Α, δεν, είναι, δεν αφορά το άρθρο 35, άρα ούτε καν μας ενδιαφέρει το επιστημονικό υπόβαθρο των εν λόγω εναλλακτικών εθνικών συστημάτων». Αυτό βέβαια θα σήμαινε ότι θα επέτρεπε η, η, Επιτροπή να υπάρχουν συστήματα τα οποία για παράδειγμα περιλαμβάνουν ένα ροζ κοντόρνι πάνω στη συσκευασία το οποίο θα σημαίνει κάτι συγκεκριμένο το οποίο όμως δεν αφορά την Επιτροπή, δεν αφορά το άρθρο 35. Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν συνάδει με το στόχο του κανονισμού. Ευχαριστώ. Η κυρία Νικολακόπουλο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Επιτροπή θα είχε προβεί σε μια αξιολόγηση του κατά πόσο ένα μέτρο πράγματι έχει αντίκτυπο στην τη λειτουργία της αγοράς, ε, ε, σε ό,τι αφορά την καταλληλότητά του ή σε ό,τι αφορά το κατά πόσο εμπίπτει στο άρθρο 35 ή όχι στο άρθρο 36 γιατί και στο πλαίσιο του άρθρου 36 προβλέπεται ότι ένα τέτοιο μέτρο έχει κοινοποιηθεί με βάση τον μηχανισμό κοινοποίηση που προβλέπεται, δηλαδή τη διαδικασία 3. Δηλαδή με βάση την οδηγία και τα τεχνικά πρότυπα. Και πράγματι, ναι, συμμετέχουν και άλλε υπηρεσίε τη Επιτροπή, ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση Γκρό, η οποία έχει αναλάβει εδώ και τον ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά δηλαδή την αξιολόγηση. Αλλά υπήρχαν και άλλες υπηρεσίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 35 και τα συστήματα δηλαδή που καλύπτονται από το άρθρο 35, ο κανονισμός προβλέπει μια δυνατότητα, δηλαδή την αρχή του ότι ένα ε, κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει δικό του εθνικό σύστημα ακόμα και αν αυτό δεν έχει επιστοποιηθεί. Έχει τη δυνατότητα το κράτο μέλο λοιπόν να θεσπίσει ένα τέτοιο εθνικό σύστημα και από εκεί και μετά προβλέπουμε κάποια κριτήρια που λέμε δεν θα πρέπει να προβαίνει σε διακρίσει, δεν θα πρέπει να ε, δημιουργεί εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των ε, ε, προϊόντων και ούτω καθεξής. Ναι, ισχύει το ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει τα κριτήρια ε, όπω αυτά προβλέπονται στο άρθρο 35 γιατί η αξιολόγηση γίνεται εκτό του 35, αλλά πάντοτε εξετάζουμε εάν μια δράση είναι απαραίτητη, εάν είναι αναλογική και προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτή την αναλογικότητα βλέπουμε εάν για παράδειγμα θα χρειάζονταν άλλα εναλλακτικά μέτρα ή όχι και επίσης ναι εξετάζουμε και την επιστημονική βάση. Η Γαλλία δηλαδή μας διέθεσε μία σειρά από ε, μελέτες και ε, εκθέσεις ε, και τεκμήρια που καταδεικνύουν ότι πρόκειται για μία δράση, για ένα μέτρο που έχει επιβάλει το οποίο λειτουργεί στην πράξη. και κατά την θέσπιση των διαφορετικών κριτηρίων για την κατάταξη δηλαδή ε, των προϊόντων ε, στο Nutri-Score, ναι, ε, βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Και επίσης η Γαλλία διοργάνωσε εδώ μια ομάδα καθοδήγησης, ένα steering group στο οποίο ε, συμμετείχαν μια σειρά από φορείς, καθηγητές πανεπιστημίου, μια σειρά από συναρμόδιοι φορείς συμμετείχαν εκεί και εμείς ε, βρεθήκαμε από την πλευρά της Επιτροπής δύο-τρεις φορές σε αυτές τις συνεδριάσεις ως παρατηρητές και κάναμε και σχόλια σε σχέση δηλαδή με το πρώτο ε, σχέδιο αυτού του συστήματος που είχε υποβάλει η Γαλλία. Και ζητήσαμε σε, αυτές, σε αυτά τα σχόλια ε, ε, μεταξύ άλλων, ε, το σύστημα αυτό να είναι εθελοντικό, να μην επιβληθεί υποχρεωτικά στι επιχειρήσει που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων. Γι' αυτό δηλαδή ζητήσαμε συγκεκριμένα από τη Γαλλία να αφαιρέσει διατάξει σε ό,τι αφορά επιβολή κυρώσεων σε τις επιχειρήσει από τον χώρο των τροφίμων. Έτσι ώστε ακριβώ η κάθε επιχείρηση του χώρου των τροφίμων να έχει δυνατότητα να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο σύστημα ή όχι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζώμα. Θα ήθελα να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα σε ό,τι αφορά τα vegetarian και τα vegan τρόφιμα. Αν κατάλαβα σωστά την Επιτροπή, μας είπε ότι δεν θεωρεί πως ε, υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναλάβει δράση. Δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να οριστούν αυτό το είδους τα τρόφιμα έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές που τα αγοράζουν πράγματι καταναλώνουν τέτοιου είδου τρόφιμα, δηλαδή φτωχογικά και βίγκα Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να οριστούν αυτού του είδου τα τρόφιμα. Okay. Ε, Κύριε ναι, θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι στην απάντηση που έδωσα δεν αναφέρθηκα στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε σε ό,τι αφορά την τεστική πράξη, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα φυτοφαγικά και τα πήγαν. Αυτό που είπα είναι ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί πως χρειάζεται να προσθέσουμε στον κατάλογο του άρθρου 36 παράγραφος 3 με βάση δηλαδή το οποίο χρειάζεται να ε, υιοθετήσουμε περαιτέρω κανόνες να προσθεθεί λοιπόν εκεί κάτι ακόμα έχουμε να ε, ε, θετήσουμε κανόνες σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα, σε ό,τι αφορά τα vegan και σε ό,τι αφορά τα reference intakes, ε, την, την, πρόληψη, πρόσληψη αναφοράς για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Αυτά είναι τα στοιχεία κατά την άποψη της Επιτροπής και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε περαιτέρω. Αλλά αν μου επιτρέπετε Πρόεδρε, επειδή τέθηκε ένα συγκεκριμένο ερώτημα από την πλευρά του κυρίου Τούρμε σε σχέση με αυτό το ζήτημα, θα μπορούσα να αναφερθώ συγκεκριμένα τώρα ε, στην ε, ε, επισήμανση των τροφίμων για φυτοφάγους, των βετζετέρια. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία, πράγματι. Η Επιτροπή εστίασε ε, τις εργασίες της, στις εκείνες οι οποίες είχαν ιεραρχηθεί ως όξος προτεραιότητα και αυτή την περίοδο υπάρχουν και περιορισμένοι πόροι με αποτέλεσμα να μην είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να δεσμευτούμε σε ό,τι αφορά μια καταληκτική προθεσμία για την υιοθέτηση των σχετικών μέτρων. Τώρα, ποια είναι η νομική κατάσταση. Οι εθελοντικές ε, πληροφορίες σε ό,τι αφορά Τέτοιε δίαιτες, τέτοια τρόφιμα δηλαδή φυτοχαϊκά και vegan, θα πρέπει να συνάδουν με τα γενικά κριτήρια, τα οποία βέβαια ενδέχεται να μην είναι αρκούντο σαφή, αλλά σε κάθε περίπτωση εμπίπτουν σε αυτέ τι υποχρεώσει. Ε, δηλαδή, θα πρέπει να είναι σαφείς οι πληροφορίες, δεν θα πρέπει να είναι αμφίσιμε, δεν θα πρέπει να παραπλανούν το καταναλωτή και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, επίση υπήρξε και νομολογία από την πλευρά του Δικαστηρίου τη Ένωση υπόθεση το Φουτάν σε σχέση με τους κανόνες τα, τους όρους σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε ε, να παράδειγμα να αναφέρεται ε, γάλα, ε, με βάση, ε, γάλα φυτικής προέλευσης, για παράδειγμα σόγιας. Εντάξει, αυτό δεν αφορά συγκεκριμένα τη χρήση του όρου vegan ή όχι, αλλά η εν λόγω νομολογία, η εν λόγω απόφαση παρέχει κάποια χρήσιμα κριτήρια στα κράτη-μέλη προκειμένου να καθορίζουν κατά πόσο τελικά η χρήση του όρου βετσετέριο φυτοβαϊκό είναι παραπλανητική ή όχι. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι ναι, υπάρχει μια αξίωση να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα για φυτοφάγους και εάν η κατάστασή μας βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κάθε περίπτωση θα ανταποκριθούμε στην ε, νομική μας υποχρέωση να λάβουμε δράση. we have... Ευχαριστώ. Μας έχουν μείνει δύο. Ένα για τις εξαιρέσεις από τον κανονισμό, τις διατάξεις παρεκκλήσεων. Μπορείτε να αναφερθείτε σχετικά, παρακαλώ. Ναι, Πρόκειται για παρεκκλήσεις ε, ε, τις οποίες αφιζητεί η κυρία Σούζεν Μέιερ. Έχει να κάνει με την εξαίρεση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή για την επισήμανση των αλκαλούχων, των αλκαλούχων ποτών σε ό,τι αφορά τα συστατικά και τα θρεπτικά συστατικά, τη, θρεπτική αξία. Και το ερώτημα είναι τι προβλέπει να κάνει η Κομισιόν, τι θα κάνει, εν περιπτώσει, το Μάρτιο του 2018, όταν θα έχουμε την έκθεση ή την πρόταση από τον κλάδο για αυτορύθμιση, για μια λύση που θα περνάει από αυτορύθμιση. Είχαμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση ε, στα πλαίσια μιας εκδήλωσης που οργάνωσε η κυρία Ζόμερ ε, πέρα από μερικές εβδομάδες με όλο τον, όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς όπου καλύψαμε πολλά ζητήματα έχουμε διαπιστώσει, η εντύπωσή μας είναι εν πάση περιπτώσει, ότι ο κλάδος ε, ε, προσπαθεί να βρει μια λύση, εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Γίνεται μια προσπάθεια να υποβληθεί μια πρόταση, παρότι υπάρχουν δυσκολίες βέβαια, υπάρχουν πολλά εκρεμή ζητήματα. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες επίσης ε, που πιστεύουμε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας. Τώρα, ε, η έκθεση της Κομισιόν βεβαίως αναφέρει σαφώς την πρόθεση εφόσον η Κομισιόν ε, θεωρήσει ότι δεν είναι ικανοποιητική πρόταση με βάση τους κανόνες για την καλύτερη νομοθεσία θα γίνει μια μελέτη αντικτύπου. Ε, αυτό είναι και μια πίεση προς τον κλάδο έτσι ώστε να υποβληθεί μια ε, λύση η οποία είναι ικανοποιητική για να αποφύγουμε τους υποχρεωτικούς κανόνες. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ε, πρώτα θα εξετάσουμε την πρόταση, την πρόταση του κλάδου. Ε, σίγουρα ε, κάποια στοιχεία που θα παίξουν ρόλο είναι ποιο είναι το επίπεδο ε, ε δέσμευσης ε, του κλάδου, ε, πόσοι δηλαδή δεσμεύονται για την προσέγγιση αυτή, διότι Προφανώς αυτό που θέλουμε είναι ε, το σύνολο του κλάδου να δεσμευθεί ε, και είμαστε βεβαίως ρυθμένοι να συζητήσουμε αυτή την πρόταση περαιτέρω με το κλάδο, αλλά και με όλους τους μπλεκόμενους φορείς, όλους τους ενδιαφερόμενους, ε, αν χρειαστεί να, προσαρμόσ, να προσαρμόσουμε τη συζήτηση αυτή, να προσ... δεν, δεν θα έρθει δηλαδή ο κλάδος με μια πρόταση την 1η Μαρτίου και η Κομισιόν μετά θα ανακοινώσει ότι είναι ικανοποιημένη ή όχι. Όχι, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εργασίες ε, κατά απόλυτα διαφανή τρόπο με όλους ε, τους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν φαίνεται να υπάρχουν ερωτήσεις. Ωραία. Θέλετε να, να προσθέσετε κάτι. Εάν δεν αφορά ε, αυτό το θέμα, παρακαλώ να κλείσουμε τις ερωτήσεις και μετά. Ε, λοιπόν, οι κανόνες για μια σειρά από θέματα, ε, εδώ δεν ε, υπάρχει χρονικός περιορισμός, ναι, είναι ένα γενικό θέμα, εδώ υπενθυμίζεται στην Κομισιόν την, ε, τις νομικές της υποχρεώσεις ε, να καλυφθούν όλα τα διάφορα ζητήματα, ιδιαίτερα την υποχρέωση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει κανόνες ε, για τις, το μέγεθος των μεριδών, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον ορισμό του φυτοφάγου και ε, τις συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών. Λοιπόν, γενικότερα να επαναλάβω κάτι που έχω πει και στο παρελθόν. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι νομικές μας υποχρεώσεις, δεν τις αμφισβητούμε, όμως από εκεί πέρα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας με βάση τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Επαναλαμβάνω, η, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιορισμοί. Σε επίπεδο πόρων ε, είναι πολύ εργασίας, ο οποίος υπάρχει και λόγω ε, απρόλεπτων εξελίξεων στο ε, στον τομέα της επισήμανσης. Ε, ε, υπάρχουν δύο-τρία άτομα τα οποία ασχολούνται μόνο με, με τις ε, προδιαγραφές για την επισήμανση και σχετική, το σχετικό νομοθέτημα, διότι ε, όπως καταλαβαίνετε γίνονται πολύ έντονε συζητήσεις και σε πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο από αυτού του θέματος. Λοιπόν, νομίζω πως απάντησα στο, στο ερώτημα για τους χορτοφάγους και για την επιλεξιμότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέγεθος των μερίδων, αυτό που είπαμε και το έχουμε συζητήσει και με τον κλάδο, προσπαθούμε να ορίσουμε τις μερίδες, ενθαρρύνουμε βεβαίως τον κλάδο ε, να αρχίσει να εργάζεται επί του θέματος αυτού, συλλέγοντας ε, ε, βέλτιστες πρακτικές ε, για το θέμα αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει και την προσπάθεια που γίνεται ε, να μπορέσει στο μέλλον η Κομισιόν ε, να έχει μια βάση. Είναι δύσκολο το έργο αυτό που έχει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποιαδήποτε πραγματογνωμοσύνη ή οποιαδήποτε ε, οι πληροφορίες από τον κλάδο είναι καλοδεχούμενες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές αναφοράς για συγκεκριμένες ομάδες όπως τα παιδιά. Ακούστε, εδώ να θυμίσω ότι αυτό, εδώ υπάρχει μια υποχρέωση. Αλλά για τις εταιρείε διατροφής μπορούν να χρησιμοποιούνται τιμές αναφορές για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία εφόσον αυτό προβλέπει του εθνικούς κανόνες. Γιατί, διότι χρειαζόμαστε επιστημονική βάση. Και η ΕΦΣΑ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τη γνωμοδότησή της για τις πληθυσμούς αναφοράς για όλους, ε, όλα τα θρεπτικά, τις θρεπτικές ουσίες. Πριν λοιπόν μιλήσουμε για συγκεκριμένες ομάδες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικαιροποιήσει ε, τις, ε, τις, τις τιμές για τον, για, πληθυσμό γενικότερα και οι τιμές αναφορές, αναφοράς για τα παιδιά ε, και τα μωρά που αναφέρονται στον 6-9 του 2013, εκεί ρυθμίζονται, εκεί που αναφερόμαστε στην διατροφή για ειδικέ ομάδες. Αυτή είναι, η, αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε και όταν ε, θα έχει ολοκληρωθεί το επιστημονικό έργο, ε, σταδιακά όταν ολοκληρώσουμε ε, τις διάφορες αναφορές ε, ε θα το κάνουμε αυτό για όλα, όλα, όλα αυτά τα μακροθρεπτικά συστατικά. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κυρία Ζόμερ, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στο πρώτο μέγεθος των μερίδων. Έχω θέσει ξανά και ξανά αυτό το ερώτημα. Πότε θα ασχοληθεί Επιτροπή με αυτό το, το, την εκπόνηση κάποιων ε, οδηγιών σε ό,τι αφορά ε, ε, το μέγεθος των μερίδων. Εδώ και πολλά χρόνια ακούω την απάντηση από την Επιτροπή δεν θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα και δεν θα ασχοληθούμε γιατί δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό. αυτό αυτή είναι η απάντηση που λαμβάνω κατά τα τελευταία χρόνια από την Γενική Διεύθυνση. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτός ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2011. Εδώ και 6 χρόνια δηλαδή βρίσκεται σε ισχύ. Και τώρα βρισκόμαστε σε ποια κατάσταση, όπου έξι ε, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δημιουργούν ένα δικό τους ε, σύστημα σε ό,τι αφορά τις ε, πληροφορίες, με βάση το μέγεθος των μερίδων και το οποίο δημιουργούν αυτές οι επιχειρήσεις μόνες τους. Και αυτό βέβαια δεν σχετίζεται με ένα γενικότερο προβληματισμό από την πλευρά των, ε, του κλάδου σε ό,τι αφορά το, τις πληροφορίες και το μέγεθος των μερίδων. Όχι. Έξι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έξι από τους global players αρχίζουν τώρα ε, να δημιουργούν ένα σύστημα σε ό,τι αφορά και τις, ε, το μέγεθος των μερίδων. Μάλλον βέβαια αντιλαμβάνεστε τι θα κάνουν εκεί. θα έχουν κάποιες μερίδες οι οποίες δεν θα είναι τόσο ρεαλιστικές. οπότε πραγματικά θα ήταν πολύ χρήσιμο αποφάσισε η Επιτροπή κάποτε ε, να θεσπίσει κάτι σε ό,τι αφορά το μέγεθο των μερίδων. Δεν θα πρέπει να αποτελέσει επιτέλου προτεραιότητα για την Επιτροπή. Θα έπρεπε να θεσπίσει δηλαδή ε, ε, κάποιε οδηγίε ό,τι αφορά τα μεγέθη μερίδων. Να αντιλαμβάνομαι ναι ότι είναι περίπλοκο ένα τέτοιο έργο και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά ναι θεωρώ πω υπάρχει ανάγκη να αναλάβει δράση. Και δεν αντιλαμβάνομαι δηλαδή γιατί εξακολουθεί να αγνοεί αυτό το ε, το ζήτημα λέγοντας απλώς ότι ε, εντάξει ο κλάδος θα, θα αναλάβει δράση εδώ. Δεν θεωρεί ότι ένας τουλάχιστον ένα τμήμα του κλάδου θα αξιοποιήσει για δικούς του σκοπούς, ιδιωτελώς αν θέλετε αυτό το κενό που υπάρχει στην νομοθεσία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Θέλετε να αντιδράσετε. Όχι. Η κυρία Κάλενμπεργκ. Κάποια ερώτηση έχετε το δικό μου ερώτημα είναι κάπως διαφορετικό από αυτό που συναδελφούζομαι. Αλλά ε, δύο ζητήματα μας έχουν απασχολήσει επανειλημμένα. Δηλαδή, ε, με συγκεκριμένη συνταγή των εισαγωγικών και αυτές που αλλάζουν δηλαδή και κατά συνέπεια η ανάγκη σήμανσης ή όχι. Ε, εμείς στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά έχουμε να κάνουμε δηλαδή με προϊόντα τα οποία οπτικά ε, δείχνουν να είναι τα ίδια αλλά αν εξεταστούν πιο προσεκτικά έχουν διαφορετικά συστατικά και τα οποία στατικά προφανώς αναφέρονται σωστά ε, στις διατροφικές χωρί χωρίς όμως να σημαίνει ότι εκ πρώτης όψεως μπορεί κανείς να διαφοροποιήσει τα δύο προϊόντα μεταξύ τους. Και η, αυτό συμβαίνει είναι ότι σε διάφορα κράτη-μέλη και σε διάφορε περιοχέ για το ίδιο προϊόν ακολουθούν διαφορετικέ συνταγέ για την παρασκευή αυτού του προϊόντο που οπτικό είναι ίδια αλλά διαφορετικό. Υπάρχει λοιπόν κάποια λύση που προετοιμάζεται έτσι ώστε να μπορεί κανεί ο καταναλωτή άμεσα και εκ πρώτη όψη να αναγνωρίζει ότι πρόκειται για διαφορετικά προϊόντα. Έτσι ώστε να γνωρίζει για παράδειγμα αν αυτό το προϊόν για παράδειγμα αφορά την Αυστρία συγκεκριμένα ή μια άλλη αγορά την Ουγγρική. Και από εκεί και μετά, μετά από το τέλος ε, των, ε, των προστώσεων που προβλέπαμε για ε, ζάχαρη, Ίσως μετά από όσα έχουμε προβλέψει για παράδειγμα τη, τη, ζάχαρη από ζαχαρότεφλα να έχουμε τώρα ε, παρασκευή προϊόντων με ισογλυκόζη περισσότερο. Και τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ ως καταναλωτής τώρα θα πρέπει πάρα πολύ προσεκτικά να εξετάζω κάθε ξεχωριστό ε, προϊόν και να βλέπω ε, περιέχει τελικά τι είδου ζάχαρη περιέχει, ή άλλη. Οπότε ε, υπάρχει κάποια υποχρέωση που προβλέπεται. Δηλαδή να αναφέρεται εκεί το είδος της με τη ζάχαρη. Και όπως είπα βέβαια ε, το ζήτημα αυτό της ε, ε, συσκευασίας και της συνταγής, δηλαδή ότι υπάρχει, υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν μια παραδοσιακή αν θέλετε συσκευασία που είναι άμεσα αναγνωρίσιμη αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα προϊόντα που είναι παρόμοια χωρίς όμως να είναι τα ίδια και αν υπάρχει ένας τρόπος για να επιληθεί αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ, όποτε θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Δυστυχώς δεν υπάρχει υποχρέωση με βάση τους υπάρχοντες κανόνες να αναφέρεται η αλλαγή ε, συνταγή, ε, τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στον κατάλογο των συστατικών. Για να ζητήσουμε από τις ε, ε εταιρείε τροφίμων να αναφέρουν ότι πρόκειται για νέα συνταγή, ε, τότε θα χρειαζόταν νέοι κανόνε. Άλλοι κανόνε στην νομοθεσία. Ε, άλλη νομοθεσία δηλαδή. Βεβαίω, ορισμένε φορέ αυτό γίνεται θελοντικά από κάποιε εταιρείε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι αλλεργίε. Ε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και με τους ασθενείς ε, ε, για τα αλλεργιογόνα. Ε, ζητείται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μια επισήμανση. Αυτό είναι, επισήμανση είναι ένα καινούριο θέμα το οποίο το εξετάζουμε και όταν θα γίνει η, ε, η αξιολόγηση των κανόνων ίσως να οδηγηθούμε προς ένα νέο πλαίσιο αλλά με βάση τους υπάρχοντες κανόνες δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε τις σημερινές μας εργασίες. Α, συγγνώμη, θέλετε να επανέλθετε σε κάποιο θέμα. Παρακαλώ. Κύριε Ζώμα, δεν έλαβα μια απάντηση και επαναλαμβάνω λοιπόν. Θα ήθελα να μου επιβεβαιώσει η Επιτροπή ότι πράγματι δεν θεωρεί ζήτημα προτεραιότητας να θεσπίσει μεγέθη μερίδων λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι έξι από τι μεγαλύτερε επιχειρήσει σε αυτό το τομέα έχουν αποφασίσει να ε, φεύγουν, αν θέλετε, δικές τους, δικά του μεγέθη μερίδων και με βάση τα οποία μεγέθη θα θεσπίσουν ένα δικό του σύστημα διατροφικών πληροφοριών. Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ουσιαστικά μια πολύ έξυπνη αλλά τελικά παρόλα αυτά παραπλάνηση του καταναλωτή. Και δεν θέλω τώρα ε, μια απάντηση με βάση το άρθρο 7. Θέλω μια απάντηση από την πλευρά της Επιτροπής ως προς το κατά πόσο θεωρεί πως η θέσπιση μεγεθών μερίδων είναι απαραίτητη ή όχι. Και αν όχι, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Γιατί στο παρελθόν μου είπε επανειλημμένα, δεν επιθυμούμε να το κάνουμε. Ακόμα και έξι λοιπόν χρόνια μετά από τη θέση εσύ του κανονισμού εξακολουθεί να έχει την ίδια άποψη. Ευχαριστώ. Ναι, όπως βλέπετε κάτι πρέπει να απαντήσετε. Ναι, ε, ετοιμαζόμουν και νωρίτερα, ε, να, ήμουν και νωρίτερα να απαντήσω. Ε, εγώ δεν διαφωνώ ακριβώ. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια νέα εξέλιξη στην αγορά, υπάρχει αυτή η νέα πρωτοβουλία. Δεν ξέρουμε βέβαια αν αυτή η πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε κάτι, θα καταλήξει κάπου. Από όσο ξέρω αυτό το πρόγραμμα είναι από συζήτηση αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα εγκριθεί. Γνωρίζουμε ότι έχει τσωματωθεί αυτή η ιδέα βεβαίως των μερίδων. Είναι κάτι το οποίο μάλιστα δεν εκτιμούν ιδιαίτερα κάποιοι από τους ε, εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων και οι καταναλωτές, δεν έχει απόψη η Κομισιόν επισήμως, αλλά έχουμε θέσει και κάποια άλλα ζητήματα εμείς που έχουν να κάνουν με την χρήση των μερίδων για την παρουσίαση αυτών των πληροφοριών. Τώρα από εκεί και πέρα ε, αντιλαμβάνομαι την εκατό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ε, είναι και νομική υποχρέωση ε, δεν λέω ότι δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουμε το θέμα ό,τι αναφέρεται στον κανονισμό ε, είναι απαραίτητο. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε το αντίθετο. Οι προτεραιότητες καθορίζονται ε, βέβαια με βάση άλλες προτεραιότητες. Ε, έτσι έχουμε εργαστεί ως τώρα. Υπάρχουν δηλαδή προτεραιότητες που καθορίζονται και με βάση συγκεκριμένε προθεσμίε που υπάρχουν, συγκεκριμένε υποχρεώσει που είχαν λάβει η Κομισιόν αντιδράσει σε ορισμένε περιπτώσει, ε, με βάση διαδικασίε διαφανεί, ε, να μπορεί ε, να απαντάει σε αιτήματα, σε έγγραφα, για πρόσβαση σε έγγραφα από πάρα, πάρα, πάρα πολλού πολίτε. Η Κομισιόν λοιπόν έχει πολλή δουλειά και ταυτόχρονα βεβαίω πρέπει να σέβεται τι νομικέ τη υποχρεώσει. Το κάνουμε, το προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ αυτό να κάνω είναι να σημειώσω αυτή τη σημερινή συζήτηση, διότι ε, αυτό που λέει η κυρία Ζόμερ είναι θεμητό ε, και είναι κάτι το οποίο θα το διαβιβάσουμε στην ιεραρχία μας ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κύριε Ζωμέρ Αν μου επιτρέπετε να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα, το οποίο ε, δεν το είχα περιλάβει στο δικό μου κατάλογο ερωτημάτων, αλλά ίσως θα μπορούσε ε, να μου το απαντήσει. Ε, για τα trans λιπαρά οξέα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια προκαταρκτική αξιολόγηση ακτικτή που είναι preliminary impact assessment και ίσω θα μπορούσε λοιπόν να μου απαντήσει η Επιτροπή στο εξή. Στην παρούσα βουλευτική θητεία θα υπάρξει μία πρόταση από την πλευρά τη επιτροπή ω προ το πώ θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των τρανσλιπαρών οξέων στα τρόφιμα. Δηλαδή, συγκεκριμένα, θα υπάρξουν οριακέ τιμέ. Γιατί διαπιστώνεται εκεί στην αξιολόγηση αντικτύπου ενδεχομένω ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν οριακέ τιμέ, όχι υποχρεωτικά επισήμανση. Οπότε το ερώτημά μου είναι, θα υπάρξει πρόταση από την Επιτροπή σε αυτή τη βουλευτική περίοδο. Thank you. Um, ναι, ευχαριστώ. Ναι, η μελέτη αντικτύπου και η δουλειά γύρω από τη μελέτη αντικτύπου είναι να εξελίξει. Ε, εμείς θεωρούμε ότι είναι εφικτό να υποβληθεί μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πριν το 2019, όπως περιπτώσει. Δηλαδή, ο σχεδιασμός μας είναι στα πλαίσια του 2018, καρδιάκια του 2018, να υποβάλουμε μια πρόταση. Τώρα, τι μορφή θα πάρει αυτή η πρόταση. Ε, θα αν θα υπάρξει μια απόφαση, αν θα πάρει τη μορφή εφαρμοστικής εκτελεστικής πράξης, ε, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, θα πρέπει να συζητηθεί. Ε, πάντως, ε, είναι εφικτό κάτι τέτοιο και ως τώρα έτσι έχουμε προγραμματίσει τις εργασίες μας. Να είναι υποβληθεί πρόταση λίγες καρδιά και αυτή τη θεία αυτή τη Επιτροπή. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο. Εάν όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνονται έτσι οι εργασίες μας για σήμερα. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στις 27 Νοεμβρίου. Καλό σας βράδυ.